dass ähm, Frau Andrula Vassilio, die vormalige Gesundheitskommissarin, Καλώς ορίζω την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, την πρώην Υπουργό, ε, Επίτροπο, με συγχωρείτε, Υγείας. Θα αναλάβει νέο χαρτοφυλάκιο, όπως την παρακάλεσε ο κύριος Μπαρόζο, δηλαδή να ασχοληθεί με τα δικά μας τα ζητήματα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσία και την νεολαία. Να υπενθυμίσω εδώ πέρα στους συναδέλφους πως έχουμε κάποιες οδηγίες για την ακρόαση, να σας, την διαβάσω, να σας διαβάσω. Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τα υποψήφια μέλη της Κομισιόν με βάση την γενική τους ικανότητα, την ε, τοποθέτησή τους όσον αφορά την Ευρώπη και την προσωπική τους ανεξαρτησία, τη γνώση τους όσον αφορά το μελλοντικό τομέα των καθηκόντων τους και την ικανότητα επικοινωνίας. Και η κυρία υποψήφια βουλευτής απάντησε σε πέντε τυποποιημένες ερωτήσεις. Τις έχετε στους ε, φακέλους σας, μπορείτε να τις ε, διαβάσετε, όπως επίσης και το βιογραφικό της σημείωμα. Θα ήθελα λοιπόν να οργανώσουμε την ακρόαση ω εξή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στην κυρία Βασιλείου για 10 λεπτά. Μετά οι συντονιστές ε, της Επιτροπής Πολιτισμού θα θέσουν από μία ερώτηση και ο κύριος Κραζόνι, ε, αντικαθίστε από τον κύριο Μέσερ Σμιτ και μετά θα ακολουθήσουν τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού. καθένας τους έχει τον χρόνο μιλίας που αναλογεί και μοιράστηκε με βάση το σύστημα αντεών της πολιτικές ομάδες. Και μετά θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που κάνουν μαζί μας την ακρόαση, καθώς πρόκειται για μια λεγόμενη συνδεδεμένη επιτροπή εδώ πέρα, στην ακρόαση αυτή, γιατί υπάρχει και επαγγελματική κατάρτιση. Και μετά θα ακούσουμε και τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας και τις ερωτήσεις τους και στο τέλος θα δώσουμε ξανά στην ε, κυρία Βασιλείου την ευκαιρία να πει κάτι στο τέλος. Ερωτήσεις και απαντήσεις ε, δεν θα κρατήσουν πάνω από πέντε λεπτά και θα έχουμε έρωτα αποκρίσεις. Δηλαδή, ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση και μετά ξανά, αν θέλετε να επανέλθετε μια δεύτερη ερώτηση, άλλο ένα λεπτό και άλλο ένα λεπτό για την τελική απάντηση της υποψηφίας επιτρόπου. Να σας πενθυμίσω πως ε, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να είναι σύντομες οι ερωτήσεις. Θα είμαι σύντομη όπως έκαναν και οι συνάδελφοι εδώ πέρα τις προηγούμενες ε, τρεις μέρες. Εάν ε, μακρηγορήσετε θα σας αφαιρώ τον λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι. ορίζω και ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Και να σας πενθυμίσω... Ναι, μετά αυτό. Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, σας δίνω τον λόγο να κάνετε τις αγωγικές παρατηρήσεις. Κυρία Πρόεδρε, έντιμα μέλη, οι ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων ενώπιον του Κοινοβουλίου αποτελούν έκφραση της δημοκρατίας και ως πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που συμμετέχω για δεύτερη φορά στη διαδικασία αυτή. Μετά τις θετικές εμπειρίες της θητείας μου ως Επίτροπος Υγείας, με ικανοποίησε ιδιαίτερα η πρόταση του Προέδρου Παρόσο να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο της παιδείας, πολιτισμού, πολυγνωσίας και νεολαίας. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο που μας φέρνει πιο κοντά στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που μας προσφέρει τα μέσα να τους βοηθήσουμε άμεσα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική εμπειρία, η οποία αποτέλεσε την πρώτη μου επαφή με το νέο μου χαρτοφυλάκιο. Πριν από μερικούς μήνες, τράβηξε την προσοχή μου μια συζήτηση μεταξύ Κυπρίων και Φιλανδών μαθητών γυμνασίων σε μια κυπριακή ραδιοφωνική εκπομπή. Μόλις είχαν ολοκληρώσει μια κοινή μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Κομένιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενθουσιασμένοι με την προσπάθεια τους, εξηγούσαν πώς τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν και να καταλάβουν όχι μόνο τις διαφορές τους, αλλά και το τι τους ενώνει. Αυτή είναι και η ουσία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ενότητα στην ποικιλομορφία. Για μένα, η συζήτηση αυτή μεταξύ των νέων μαθητών ήταν εξαιρετικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχουμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σας για τις βασικές μου προτεραιότητες. Να ενισχύσουμε την επιμόρφωση των πολιτών και να διευρύνουμε την πρόσβαση στην παιδεία και την εκπαίδευση με έμφαση στις, εξειδικεύσει που αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες της σημερινής οικονομίας, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης. Να αυξήσουμε τις ευκαιρίες και την κινητικότητα της νεολαίας μας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα προάγει τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα σε ατομικό επίπεδο, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. In Europe, Madam President... Κυρία Πρόεδρε, αν η Ευρώπη θέλει να πετύχει στον ανταγωνισμό μέσα στη νέα παγκόσμια οικονομία, τότε πρέπει να δώσουμε νέες ευκαιρίες για αριστεία, για έρευνα και για καινοτομία. Πρέπει να εξοπλίσουμε τους νέους μας με υψηλά προσόντα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο μέλλον. Η ανώτερη εκπαίδευση είναι ζωτική σημασία παρά τα πραγματικά, την πραγματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τη διαδικασία της Βολόνιας, ε, τα πανεπιστήμια μας ακόμα δεν ανήκουν στα καλύτερα στον κόσμο αρκετά όσο θα έπρεπε. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση όπως και η εκπαίδευση για τους ενήλικες χρειάζονται εξυγχρονισμό. Πρέπει να ενισχύσουμε την κατάρτιση των διδασκόντων επίσης. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε να μοιράσουμε καλύτερα στον κόσμο τα κέρδη από τη νέα οικονομία αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την ύφεση και αν θέλουμε να πετύχουμε μια περισσότερο ευφυή, πιο πράσινη κοινωνία της γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βοηθήσουμε με δραστήριο τρόπο τον ένα στους έξι νέους οι οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο πριν το ολοκληρώσουν. Τον ένα στους πέντε 15 που δεν είναι σε θέση να διαβάσουν καλά-καλά και τα 80 εκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν με πολύ χαμηλά και βασικά προσόντα. Χρειάζονται περισσότερε επενδύσει στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη όπου όλοι να διαθέτουν τα προσόντα να υποφεληθούν από τι νέε ευκαιρίε μετά την κρίση η δικιά σας στήριξη για να βοηθήσετε με πόρους την Ευρώπη όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτική σημασία. Γι' αυτό χρειάζεται να διασφαλίσουμε και τη στήριξη των εθνικών κυβερνήσεων, των περιφερειακών αρχών και του ιδιωτικού τομέα. Αποτελεί και αυτό μια σημαντική πρόκληση για όλους μας. Η προτινόμενη στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδει ένα ρόλο κλειδί στην εκπαίδευση και την κατάρτιση που αποτελούν κινητήρια δύναμη, ένα μοχλό για υψηλότερα προσόντα και δεξιοτεχνίες που θα τροφοδοτήσουν μια αηφόρο βασισμένη στη γνώση ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θέλω επίση, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία, όσον αφορά τι δράσει Μαρή Κιουρκέ, το Erasmus Mondus, το πρόγραμμα Erasmus να φροντίσω να συνεισφέρουν σε μια ξεχρονισμένη ανώτατη εκπαίδευση και να βοηθήσουν η Ευρώπη να γίνει πιο ελκυστική για σπουδέ και έρευνα. Θα σα πω πώ σκοπεύω να βοηθήσω το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία προκειμένου να αποτελέσει τη σημεοφόρο τη Ευρωπαϊκή κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση. Οι δράσει Marie Curie θα ενισχύσουν τι προσπάθειέ μα προκειμένου να φέρουμε πιο κοντά του ευρωπαϊκού χώρου τη ανώτερη εκπαίδευση και έρευνα, έτσι ώστε η γνώση και οι ερευνητέ, οι φοιτητέ και το προσωπικό που φροντίζουν για να δημιουργηθεί αυτή η γνώση να μπορούν να κινούνται ελεύθερα ε, στα σύνορά έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αριστεία στην έρευνα και στην εκπαίδευση, που θα οδηγήσουν με τη σειρά του σε καινοτομία. Μια άλλη μεγάλη προτεραιότητα για μας και σημαντική είναι να γενικεύσουμε και να επεκτείνουμε την κινητικότητα όσον αφορά την μάθηση μέσω του προγράμματος Νεολαία σε κίνηση. Όπως δείχνουν και τα προγράμματά μας, πιστεύουμε ότι η κινητικότητα μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά σε βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων όλων των νέων μας. Όπως επίσης ανοίγουν και το πνεύμα μας σε, νέες, πολιτισμούς και νέα ηθικέθημα. Στόχος μας είναι λοιπόν όλοι οι νέοι στην Ευρώπη να μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες και άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της μάθησης, όπως είναι οι διδάσκοντες, και αυτοί να μπορέσουν να επωφεληθούν από την κινητικότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα. Στόχος μου είναι λοιπόν να φροντίσω γι' αυτό το μελλοντικό πλαίσιο όσον αφορά την νεολαία σε κίνηση το καλοκαίρι που θα μας έρθει. Όπως ε, έχει θέσει και στις πολιτικές του κατευθυντήρες γραμμές ο πρόεδρος Βαρόσο, πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία η οποία θα είναι αποφασιστική σημασία για την πολιτιστική ποικιλομορφία, τον πολιτιστικό διάλογο και την πολυγλωσία. Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ μέσα από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό να προωθήσω αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η Ευρώπη, αλλά να στηρίξω επίσης και τη δημιουργία και την καινοτομία. Γι' αυτό πρέπει να ελευθερώσουμε όλο το δυναμικό που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Κλάδος Πολιτισμού και Δημιουργίας. Θα δοκιμάσουμε μια πράσινη βίβλο να εντοπίσω τις ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις οι οποίες βοηθούν τους Ευρωπαίους δημιουργούς να εκφραστούν καλύτερα. Επίσης, μόλις είναι έτοιμο το νέο σώμα των επιτρόπων, να υποβάλω μία πρόταση για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ε, σήμα κληρονομιάς πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Πιστεύω πράγματι ότι είναι κάτι συμβολικό, το οποίο όμως θα μας βοηθήσει πολύ, διότι θα δώσει μεγαλύτερη προβολή στους χώρους εκείνους που δίνουν ε, πνοή και ζωή στα ιδεώδη της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα οικονομικό ή πολιτικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει ως στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει την πολιτιστική μας ποικιλομορφία και τις αξίες μας. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πολύ που ο πρόεδρος συμπλήρωσε το χαρτοφυλάκιο αυτό με το πρόγραμμα Media. Ο κινηματογράφος είναι και πρέπει να παραμείνει ένα σημαντικό μέσο έκφρασης για την ευρωπαϊκή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το πρόγραμμα Media λοιπόν συγκεκριμενοποιεί και αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή δέσμευση που είναι πολύ ισχυρή και όχι βέβαια σημερινή σε αυτό το τομέα. Η κοινοτική δράση πρέπει να βοηθήσει να φανεί η πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, να βοηθήσει επίσης για ένα ανταγωνιστικό κλάδο στην διεθνή σκηνή, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Αυτή είναι η πρόκλησή μας. Γι' αυτό θα βασιστώ στις παλιότερες επιτυχίες μας και θα δώσω ιδιαίτερη σημασία στον αντίκτυπο που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον κινηματογράφο. Επίσης θα είμαι ιδιαίτερα προσεκτική προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διανομή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου διεθνώς. Στόχος μας πρέπει να είναι να προωθήσουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία και την πολυγλωσία και αυτό μέσω όλων των εξωτερικών μας πολιτικών. Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά με την πολυμορφία που την διακρίνει και που χαρακτηρίζει την Ευρώπη πρέπει να μεταφέρει τη φωνή μας και τα οράματά μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Και γι' αυτό η σύμβαση της UNESCO μας προσφέρει μια στέρεα νομική βάση και έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ προκειμένου να εισαγάγουμε πολιτιστικές προτεραιότητες και σε άλλες πολιτικές. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των συγγραφέων. Εδώ θέλουμε να διασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα από τη μια μεριά σωστέ, καλέ αμοιβέ για του δημιουργού, κάτι το που είναι ζωτική σημασία για τη δημιουργία και την πολιτιστική πολυμορφία, και από την άλλη μεριά να έχουμε μια ευρύτερη πρόσβαση του κόσμου στον πολιτισμό. Επ' αυτού θέλω να συνεργαστώ στενά μαζί με τους άλλους επιτρόπους συναδέρφους μου πάνω σε μια νέα ψηφιακή ατζέντα η οποία να σέβεται την ισορροπία αυτή. Τέλος θα προσπαθήσω βέβαια να στηρίξω την πολυγλωσία, την γλωσσική πολυμορφία, την εκμάθηση ξένων γλωσσών που αποτελούν ένα μέσο για περισσότερη αποσχόληση και επίσης αποτελούν και μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της κληρονομιάς που θα μεταφέρουμε στους επόμενους. Με συγχωρείτε, δεν είμαι πολύ γενική, αλλά πρέπει να σας διακόψω γιατί πέρασαν τα δέκα λεπτά σας. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, της ε, Επιτροπής να λάβουν λόγο. Θα είμαι ακόμη πιο ε, αυστηρή. Ο κύριος Κουρία, λοιπόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την κυρία Βασιλείου και θα ήθελα να εμβαθύνω σε ένα σημείο από αυτά που μας είπατε για να καταλάβω καλύτερα περί τίνος πρόκειται με το νέο αυτό πρόγραμμα για το οποίο μας μιλήσατε, η κινητικότητα των νέων και πώς μπορούμε να συντονιστούμε με το πολιετές πρόγραμμα που έχουμε. Η νεότητα σε δράση βοήθησε πάρα πολύ αυτό σε ανταλλαγή, στην ανάπτυξη της κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη. Να δούμε τι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για να γίνει πιο αποτελεσματικό και καλύτερο το πρόγραμμα αυτό με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντικής Δράσης με προοπτική το 2011 που όπως ξέρετε είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Ευχαριστώ κυρία Βασιλείου. Ναι, το πρόγραμμα νεολαία σε κίνηση είναι κάτι το οποίο θα αγκαλιάσουμε και θα απλοποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο, γιατί μελετώντας αυτό το χαρτοφυλάκιο, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι τα πάρα πολλά προγράμματα και η ποικιλομορφία των όρων που χρησιμοποιούμε και ίσως να δημιουργούν κάποια σύγχυση στους νέους και στους λαούς μας. Ειδικά στους νέους που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα προγράμματα. Οπότε, όταν μελετήσαμε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, την οποία οπωσδήποτε θα προετοιμάσουμε συνεργασία μαζί σας και λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας ιδέες. Ξεκινάμε με την, με την κινητικότητα της νεολαίας από τους μαθητές μέχρι τους ερευνητές, ε, από τον πολιτισμό μέχρι τον αθλητισμό. Και βέβαια ε, το ζήτημα του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θεωρούμε πως ο εθελοντισμός βοηθάει τους νέους ε, να αποκτήσουν καλύτερες εμπειρίες ε, και να μάθουν περισσότερα πράγματα στην ζωή. Οπότε ουσιαστικά αυτή θα είναι η πολιτική μας για την κινητικότητα και τον νεολαία για το μόνο. Και όχι μόνο. Και λέω όχι μόνο γιατί πρέπει να λέω υπόψη και τους ενήλικες, όχι μόνο τους νέους. Γιατί όταν μιλάμε για διαβίου μάθηση, προφανώς δεν σταματάει όταν ε, αποφυτίσει κανείς ή όταν βρει δουλειά. Πρέπει να συνεχίζεται γιατί οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Και πρέπει να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους αυτή τη δυνατότητα να μαθαίνουν, να αποκτούν εμπειρίες, ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση, μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να επανέλθετε κυρία Σκουρία με άλλη ερώτηση. Μία διευκρίνηση μόνο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη και τους μαθητές και τους φοιτητές και πέραν του πανεπιστημίου αυτούς που θέλουν να μπουν στον χώρο εργασίας. Πολλές γενιές λοιπόν για να εξασφαλιστεί μια κοινή ευαισθησία. Γι' αυτό μιλάμε, κατάλαβα καλά. Well, it's it's it's a chain. Είναι μια αλυσίδα Του ξεκινάει από το δημοτικό και πριν από αυτό και τελειώνει όταν κάποιος βρίσκει κάποια απασχόληση και πιο μετά. Οπότε θέλουμε να διευρύνουμε το φάσμα σε όλο το μήκος αυτό της ε, αλυσίδας. Γιατί βεβαίως δεν μπορεί κάποιοι κρίκοι να είναι πιο αδύναμοι από τους άλλους. Και με την ε, πράσινη βίβλο για την κινητικότητα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εμπόδια για την κινητικότητα και να τα αντιμετωπίσουμε για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους να εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα. Σας ευχαριστώ κυρία Χάνιμπολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Βασιλείου. Η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, ζητούν ε, εδώ και χρόνια από την ε, Κομισιόν να βάλει τα συμφέροντα των πολιτών στο κέντρο της στρατηγικής 2020. Ε, ειδικά στους δύσκολους καιρούς, τους οποίους αναφέρατε. Και θέλω να σε ρωτήσω, εάν συμφωνείτε πως η νέα στρατηγική του 2020 πρέπει να περιέχει και μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, που εγώ τουλάχιστον νομίζω και θέλω να μάθω τη δική σας άποψη, ότι θα είναι πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και της ανισότητας. Και εάν σε αυτό το πλαίσιο θα ε, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε συγκεκριμένες ιδέες για την ενίσχυση της ε, κοινωνικής ένταξης, όχι μόνο μέσω της εκπαίδευσης, την οποία αναφέρατε, και πώς θεωρείτε ότι μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο η καλύτερη εκπαίδευση για κατάρτιση. Η κυρία Βασιλείου, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι βεβαίως ναι. Είμαι υπέρ της κοινωνικής ένταξης όλων και όταν μιλάμε για τις ευκαιρίες που πρέπει να δίνουμε στους νέους και στους ανθρώπους γενικά, πρέπει να δώσουμε βάρος στους ανθρώπους που προέρχονται από φτώχειες οικογένειες ή από ομάδες οι οποίες ε, έχουν κάποια μειονεκτήματα, είτε μιλάμε για παιδιά μεταναστών ή παιδιά γονιών ε, που δεν έχουν κάποια μόρφωση, κάποια εκπαίδευση. Οπότε πρέπει να συμπεριλάβουμε τους πάντες. Και για να γίνει αυτό δεν φτάνει να μιλάμε μόνο για την επίσημη τυπική εκπαίδευση, η οποία βεβαίως είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες ε, μορφές εκπαίδευσης, άτυπη, ανεπίσημη αν θέλετε, εκπαίδευση και βεβαίως ε, να αυξήσουμε και τις γλωσσικές τους ε, ικανότητες. Και αυτό είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο απασχολησιμότητας και πρέπει αφενός να προσπαθήσουμε να ταιριάξουν από τη μία οι δεξιότητες τους ε, με τις δουλειές οι οποίες υπάρχουν. Εάν μου επιτρέπετε λοιπόν μια συμπληρωματική ερώτηση, να δούμε λίγο την κοινωνική διάσταση, την ανεργία και το πώς τα μέτρα τα οποία αναφέρατε θα οδηγήσουν σε θέσεις απασχόλησης. Γιατί κατά βάση όταν μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό η αιτία είναι περισσότερο οποιαδήποτε άλλη ανεργία. Η κυρία Βασιλείου, σύμφωνα με τις μελέτες μας, γύρω στο 50% των αποφύτων του Πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι. Γιατί? Πρέπει να βρούμε γιατί. Και σε κάποιες χώρες είναι ακόμη υψηλότερο το ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε και να συνδέσουμε τις δεξιότητες και τη γνώση με την απασχόληση. Δεν έχει νόημα να έχουμε αποφύτους που δεν βρίσκουν δουλειά. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς. Οπότε θα κάνουμε μία μελέτη και θα δούμε από αυτήν τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες για τους ανθρώπους να έχουν καλύτερη κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση. Κοίτα, προερχόμενοι από τον τομέα της υγείας, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως έχουμε έλλειψη γιατρών, νοσοκόμων, ειδικών και νομίζω πως πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να κατευθυνθούν προς αυτά τα επαγγέλματα γιατί θα βρουν σίγουρα δουλειά. Σας ευχαριστώ. Κατόπιν ο κύριος Στάκουλα. Κύριε Υποψήφα Επιτροπή, καταρχήν σας συγχαίρω για την άρεστη παρουσίαση που μας κάνατε. Στα αποτελέσματα της πίσας βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στα, το τι ισχύει σε μία χώρα και τι ισχύει άλλη. Ερωτώ, θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία θα πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά την εκπαίδευση και πώς προτείνεται αυτό να γίνει προς αμοιβαίο όφελος της κάθε χώρας μέλος ανταλλάσσοντας εμπειρίες σε διάφορους τομείς. Απάντηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο εναρμονισμένο σύστημα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις χώρε μέλη να ανταλλάσσουν τις καλύτερες εμπειρίες τους και να του υποστηρίζουμε σε αυτό. Και αυτό το κάνουμε εδώ και κάμποσα χρόνια. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα το τέλειο, αλλά αυτή είναι η μόνη λύση η συνεργασία και η ανταλλαγή των άριστων μεθόδων. Το να ορίσουμε δείκτες, παραδείγματος χάρη, δεν είναι σαν να προσπαθούμε να ξεμπροστιάσουμε κάποια χώρα. Τους δίνουμε μια κατευθυντήρια, μια κατεύθυνση. Ποια είναι τα ασθενή σημεία, πώς μπορούν να τα βελτιώσουν, διότι τα ασθενή και τα ισχυρά σημεία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πρέπει να δούμε λοιπόν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ποια είναι τα ασθενή σημεία. Η πρόεδρος διακόπτη. Ναι, συγγνώμη, ήταν... Ναι, ήταν η πρώτη ερώτηση. Έχετε, έχετε ακόμη χρόνο. Ναι, ήταν η πρώτη ερώτηση. Συγγνώμη, έχετε δύο λεπτά, έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Η υποψήφη επίτροπο συνεχίζει. Ξέρω, όταν έγινε η τελευταία μεγάλη διεύρυνση, είχαμε πάρα πολλά κενά και στην εκπαίδευση και σε πολλούς άλλους τομείς. Ήταν φυσικό αυτό. Προσπαθούσαμε λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα στις νέες χωρισμένοι να βελτιωθούν τα συστήματά τους και έχουμε καλά παραδείγματα. Η Σλοβενία, Φερρυπίν, που είχε ένα πολύ ασθενές εκπαιδευτικό σύστημα, αξιοποίησε τα προγράμματά μας, τη βοήθειά μας και τώρα βλέπουμε ότι στη χώρα αυτή έχει σημειωθεί μια μεγάλη βελτίωση. Αυτή είναι η λύση. Να δούμε τι έχουν κάνει οι άλλε χώρε και να προσπαθούμε ο καθένα να βελτιώνει το σύστημά του. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. So, I don't think that anyone... Νομίζω ότι κανένας εδώ μέσα δεν θα αμφισβητήσει το σημαντικό ρόλο γι' αυτό που είπατε. Όπως επίσης και η εκπαίδευση των διδασκόντων δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί. Θα επενδύσετε στην εκπαίδευση των διδασκόντων στην Ευρώπη. Απάντηση. Καταρχήν έχω να σας πω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι διδάσκοντες, η δεξότητα τους, η εκπαίδευση τους, τα προσόντα τους και οι διδακτικές μέθοδοι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ίσως είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των μαθητών και των σπουδαστών. Και όλοι έχουμε προσωπικές εμπειρίε από αυτό. Διάβαζα ένα άρθρο χθε το βράδυ για τις νέες τεχνολογίες και είναι καταπληκτικό. Αντί να έχουμε ε, κενά γενεών, τώρα έχουμε κενά κάθε πέντε χρόνια λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία πώς οι διδάσκοντες θα τα φέρουν βόλτα με όλες αυτές τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στη διδασκαλία γλωσσών κλπ. Αν δεν τους εκπαιδεύουμε συνεχώς. Η αρχική εκπαίδευση είναι καλή, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση, η διαρκής εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική. Και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Πρέπει να τους δώσουμε ειδικά μαθήματα, γιατί μπαίνουν στην εκπαίδευση και δεν ξέρουν, παραδείγματος χάρη, ε, δεν γνωρίζουν πολλά για την παιδαγωγική διάσταση. Πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτό. Σας ευχαριστώ η κυρία Μπεναράμπ Ατού. Bonjour, euh, Madame Vassiliou, et bienvenue. Καλημέρα κυρία Βασιλείου, καλώς ορίσατε. 25% των 15 ετών στην Ευρώπη δεν είναι στη θέση να διαβάζουν πάρα πολύ καλά. Και σήμερα στην Ευρώπη βρισκόμαστε κάτω από το πλαίσιο αναφοράς. 6 εκατομμύρια νέων κάθε χρόνο εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα. Το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας για να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός και να έχουμε πρόσβαση των ατόμων με δυσκολίες νέων και λιγότερων νέων στις βασικές γνώσεις. Και στην προοπτική αυτή και λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Συνθήκης Λισαβόνας δεσμεύεστε να προτείνετε στο Συμβούλιο την αύξηση του προπολογισμού για τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. κυρία Βασιλείου θα απαντήσει. Ξέρω ότι η έκθεση του περσμένου Νοεμβρίου δείχνει σαφώς ότι δεν πετύχαμε τους στόχους που είχαμε ορίσει για το 2010. Πρέπει όμως να επιμείνουμε. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να επιμείνουμε στη βελτίωση της ποιότητας των επιδόσεων των παιδιών μας, διότι όλοι συμφωνούμε ότι αν τα παιδιά δεν έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται στη ζωή, δεν θα έχουν επιτυχία. Πρέπει λοιπόν να το τονίζουμε αυτό, την εκπαίδευση τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Γιατί όπως είπα και πριν, τα παιδιά τους τραβάει πάρα πολύ η νέα τεχνολογία. Και πιθανότητα ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή ο γλωσσικός, ο αναγνωστικός μάλλον αλφαβητισμός είναι αυτό που αναφέρεται, είναι ότι τα παιδιά παραπέζουν πολύ με τα video games. Αλλά είναι φυσιολογικό αυτό, τα παιδιά τους τραβάει αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ενδιαφερθούν και για τη λογοτεχνία, την ανάγνωση, άρα να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Αλλά και με την κινητικότητα και τα σχετικά προγράμματα θα πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά να ενδιαφέρονται περισσότερο στο να συνεργάζονται με άλλα παιδιά από χώρες που τα πάνε καλύτερα, που έχουν καλύτερες επιδόσεις. Ανταλλαγές λοιπόν. Κατάρτιση και προσόντα των διδασκόντων. Επίσης σημαντικό και αυτό. Σε αυτό θα δώσω έμφαση για να πετύχουμε τους νέους στόχους, τους πιο φιλόδοξους στόχους για το 2020 που θα σας τους παρουσιάσουμε φέτος. Συμπληρωματική ερώτηση. Δεν απαντήσατε στο ερώτημα κατά πόσο να δεσμεύεται να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τα πρόγραμματα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Απάντηση. Φυσικά δεσμεύομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ να βελτιωθεί ο προπολογισμό. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εγώ θα δώσω μάχες για ένα σωστό προπολογισμό. Αλλά χρειάζομαι την υποστήριξή σας, την υποστήριξη των Υπουργών και πρέπει στο μέλλον να στηριζόμαστε και σε άλλους εταίρους, τοπικές και περιφερειακές αρχές, να επενδύουν περισσότερα στους τομείς αυτούς και στη βιομηχανία. Αν συνδέσουμε την, τις γνώσεις, την εκμάθηση με τη βιομηχανία, τότε ο τομέας αυτός θα ενδιαφερθεί περισσότερο, θα επενδύσει περισσότερο και αυτός. Η κυρία Μακλάκιν. Καλώς ήρθατε. Κύριε Βασιλείου. Το δικό μου το ερώτημα αφορά τις νέες αρμοδιότητες στον αθλητισμό μετά τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Πώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε μια πολιτική που θα αφορά τον μαζικό αθλητισμό και εξάλλου αυτή είναι η καλύτερη πολιτική για να βελτιωθεί ο αθλητισμός και να καταπολεμηθεί και η παχυσαρκία και να αυξηθεί η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να αυξήσετε τον μαζικό αθλητισμό αλλά και όσον αφορά τον επαγγελματισμό ε, αθλητισμό που δυστυχώς επικεντρώνεται κυρίως η νομοθεσία και ειδικά στο ποδόσφαιρο πρέπει να σκεφτούμε και άλλα μειονοτικά αθλήματα και το πώς θα έχουμε μια πολιτική για τον αθλητισμό που θα αφορά όλα τα αθλήματα και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Κύριε Βασιλείου, Λυπούμε για το ότι δεν μπόρεσα να τελειώσω τις αρχικές μου παρατηρήσεις για το, το τελευταίο κομμάτι αφορούσε τον αθλητισμό. Αλλά πρέπει να τονίσω πως για εμένα ο αθλητισμός είναι πλέον έκτημα και μπορεί να ωφελήσει τους πάντες. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση του αθλητισμού, αλλά και η κοινωνική. Και ο μαζικός αθλητισμός είναι η θα έπρεπε να είναι βάση της πολιτικής μας. Γιατί ωφελεί την υγεία και το ξέρω γιατί πρόσφατα διοργάνωσα ένα ειδικό συνέδριο για την νεολαία και την υγεία και ο αθλητισμός. Η σωματική δραστηριότητα γενικά είναι πολύ σημαντικός τομέας και επίσης για να κινητοποιήσουμε όλους τους νέους που υπάρχουν, ο καλύτερος τρόπος είναι ο αθλητισμός. Ο εθελοντισμός μέσω του αθλητισμού είναι ο καλύτερος τρόπος. Και να σας πω και μια προσωπική μου εμπειρία. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το Special Olympics στην Κύπρο πριν από λίγα χρόνια. Είχα πάει με την εθνική ομάδα σε δύο διεθνείς ε, συναντήσεις και πανευρωπαϊκούς αγώνες. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το όφελος που είχαν αυτά τα παιδιά από τον αθλητισμό. Και κάποια από αυτά τα παιδιά τώρα είναι πλέον ανεξάρτητα. Εργάζονται και πήραν τη ζωή τους στα χέρια τους. Οπότε ο αθλητισμός είναι πραγματικά ε, βάση, η βάση για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Κυρία Μακλάρκιν, θέλει συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Σας ευχαριστώ για την έμφαση που δίνει στον αθλητισμό. Συμφωνώ πλήρως. Ελπίζω να παίξει και σημαντικό ρόλο στο χαρτοφυλακία σας. Είστε φίλαθλος ίδια και τι, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την διοίκηση του αθλητισμού και το πώς λειτουργεί αυτή και πώς θα εργαστεί το κομμάτι αυτό εντός της γενικής σας διεύθυνσης. Ε, η κυρία Βασιλείου. Ναι, να είμαι ειλικρινή. Είμαι φιλαθλό, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλο. Ε, μπορεί να γίνω στο μέλλον, δεν με πειράζει. Γιατί ο εγγονό μου ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον αθλητισμό. Ο πατέρα μου επίση πάρα πολύ για το ποδόσφαιρο. Οπότε έχω ερεθίσματα, αλλά ο αθλητισμό για μένα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι το τέννη, το μπάσκετ, το βόλεϊ, η κολύμβηση. Είμαι καλή κολυμβήτρια ε, επί τη ευκαιρία προέρχομαι και από νησί. Οπότε ασχολούμαι πάρα πολύ με τον αθλητισμό όταν ήμουν νέα. Εξακολουθώ να γυμνάζομαι. Οπότε ο αθλητισμός θα αποτελέσει για μένα ένα σημείο στο οποίο θα δώσω έμβαση και μαθαίνω κιόλα αρκετά καλά. Ό,τι δεν ξέρω θα το μάθω από τους εφισταμένους μου στις ε, υπηρεσίες μου και με τη βοήθειά τους είμαι σίγουρη πώς θα είμαι σε θέση να προωθήσω και αυτό το κομμάτι των αρμοδιοτήτων μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά είναι εδώ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, εδώ είμαι. Ευχαριστώ κυρία Βασιλείου. Καλώς ήρθατε. Πολιτισμός, εκπαίδευση είναι πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν και στην καρδιά των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα μάλιστα ίσως καλύτερα γιατί όπως είπατε κι εσείς και υπογραμμίσατε ότι καταρχήν ξεκινήσαμε με μια οικονομική Ευρώπη. Έχετε δίκιο το ευρωπαϊκό σχέδιο όμως δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτό διότι ο πολιτιστικός χώρος είναι ένα του για την Ευρώπη η ποικιλομορφία είναι πλούτος, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα χάσμα πολύ όλο μεγαλώνει μεταξύ πλουσίων και φτωχών και αυτό ισχύει και στον πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξέρω εσείς πώς θα ενισχύσετε την μη επαγγελματική κατάρτιση που ο στόχο δεν θα έχει δηλαδή τις ανάγκες της αγοράς. Μας μιλήσατε για το πρόγραμμα νεολαία σε κίνηση. Δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε απόλυτα ότι είπατε γι' αυτό. Πρέπει να ολοκληρώσετε κυρία Βεριζιά ή κυρία Βασιλείου. Ναι, η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί μέρος της αλυσίδας της διαδικασίας μάθησης. Είναι ένας κρίκος της αλυσίδας αυτής. Από τους καλύτερους επαγγελματίες ε, ξέρουμε ότι έρχονται από πολύ σημαντικά Ινστιτούτα επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Όμως, ό,τι έχουμε κάνει με την ανώτερη εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας της Μπολόνια δηλαδή, δεν μας βοήθησε στον τομέα της επαγγελματική κατάρτισης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας και να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες. Πρέπει να ενισχύσουμε τα αισθητούτα επαγγελματική κατάρτισης και πρέπει να υπογραμμίσουμε το θέμα της ποιότητας της κινητικότητας, των δυνατοτήτων απασχόλησης που προσφέρονται και να δούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να συγκλίνουν τα διάφορα συστήματα για να αναγνωρίζονται τα πτυχία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί και η δυνατότητα που έχουν τα, κράτη-μέλη να προσφέρουν κινητικότητα σε αυτό το τομέα. Έπειτα, όσον αφορά το πρόγραμμα νεολαία σε κίνηση, η επαγγελματική κατάρτιση είναι μέρος των προσπαθειών μας, διότι εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στις ε, δεξιότητες, στα προσόντα που τα παίρνει κανείς και από την εκπαίδευση και από την επαγγελματική κατάρτιση. Η κυρία Βερζιά, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Μάλλον δεν με καταλάβατε καλά. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ακριβώς εμείς έχουμε μανία με την επαγγελματική κατάρτιση και τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση που εξετάσαμε όσον αφορά τη σχέση πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι το χάσμα που υπάρχει όσον αφορά τις πολιτιστικές δυνατότητες, κοινωνικές επιστήμες. Πράγματα τα οποία από ό,τι φαίνεται μένουν αποκλειστικά σε μία ελίτ και όλο και περισσότερος κόσμος μένει εκτός. Παράδειγμα, το Ευρωπαίανα είναι ένα καλό παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε. Δείχνει δηλαδή ότι την πολιτιστική Ευρώπη πρέπει επίσης να τη χτίσουμε και να της δώσουμε προτερότητα. Η κυρία Βασιλείου. να μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο. Και χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη συνεργασία. Να ενισχύσουμε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά ώστε να ανταποκρίνεται και σε άλλες προκλήσεις που έχουμε. Προκειμένου πάντως να το πετύχουμε αυτό, Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν και εκείνα. Πρέπει να έχουν καλύτερες προδιαγραφές για την ψηφιακή μας κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που θα προωθήσουμε εγώ και συναδελφοί μου επίτροποι, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει συντονισμένα να δράσει στον τομέα αυτό. Είμαι σίγουρη ότι η νέα Επιτροπή και οι νέοι Επίτροποι θα συνεργαστούν πολύ καλά μεταξύ τους για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστούμε. Μέσερ Σμιτ τώρα, κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επανέλθω σε κάποια θέματα που αναφέρατε και εσείς εισαγωγικά. Αναφερθήκατε στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Ξέρω τι έχει γίνει στον τομέα του πολιτισμού με τον προπολογισμό τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία με εκπλήσουν. Χρηματοδοτήσαμε ορισμένα πράγματα, γκολ στην Πορτογαλία ή στη Σουηδία ή ένα θέατρο για μαριονέτες στις βαλτικές χώρες. Εμένα όλα αυτά με μπερδεύουν, γιατί βλέπω πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, τουλάχιστον διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Τελικά, μήπως πρόκειται για χάσιμο χρημάτων, για σπατάλη, έτσι θα φτιάξουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Η κυρία Βασιλείου. Κοιτάξτε, οι υποδομές για τον πολιτισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι αναγκαίο. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι ο στόχος των προγραμμάτων μας. Έχουμε άλλα προγράμματα που έχουν αναλάβει άλλες γενικές διευθύνσεις, περιφερειακά προγράμματα για παράδειγμα που βοηθούν και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη επωφελούνται από τα προγράμματα αυτά για να ενισχύσουν τέτοιες υποδομές. Αυτό όμως που εμάς μας ενδιαφέρει, τη δικιά μας γενική διεύθυνση, είναι να ενισχύσουμε την ανθρώπινη πλευρά του πολιτισμού, να δώσουμε δηλαδή δυνατότητες στους καλλιτέχνες μας να δημιουργούν, να ανταλλάσσουν επίσης ιδέες και να εμπνέονται από δημιουργίες άλλων χωρών. Τέτοια προγράμματα εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ανέφερα προηγουμένως το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θέλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσει περισσότερο νόημα στην αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη των πολιτών μας. Όλοι αυτοί οι πολιτιστικοί χώροι οι οποίοι θα βρεθούν κάτω από αυτό το σήμα καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει. Ο κόσμος θα μάθει καλύτερα την ιστορία μας, τις πολιτιστικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας. Είναι ένα είδος προγράμματος που εμείς θα προωθήσουμε και θα προωθήσει και αυτό με τη σειρά του την πολυμορφία την πολιτιστική στην Ευρώπη. Ένας άλλος τρόπος είναι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Άκουσα τι γίνεται με τις φετινές πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, το είναι για παράδειγμα, όπου παραδοσιακά ήταν μια βιομηχανική περιοχή. Τώρα όμως που η πόλη αυτή είναι ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα, η πόλη αυτή θα πάρει ένα άλλο χρώμα, θα είναι ένα πολιτιστικό κέντρο. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ. Θέλω να βεβαιωθώ ότι σας κατάλαβα καλά. Γιατί αν δείτε τι έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια, με τα χρήματα του φορολογούμενου. Εσείς πιστεύετε ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν καλά. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή τη ότι χρησιμοποίησε καλά τα χρήματα αυτά σε, στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι σας καταλαβαίνω καλά σε αυτό που μας λέτε. Γιατί στα κράτη-μέλη πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί εκλογείς, πολλοί πολίτες, άντρες και γυναίκες που πιστεύουν ότι είναι πολύ περίεργο να βλέπουμε προγράμματα με τεράστια ποσά, ενώ θα μπορούσαμε τα χρήματα αυτά να τα είχαμε χρησιμοποιήσει για την έρευνα, για παράδειγμα, για άλλα πράγματα. Θέλω λοιπόν να ξέρω ακριβώς ποια είναι η θέση σας. Συμφωνείτε για το ότι σπαταλήθηκαν χρήματα ή όχι. Βασιλείου. Η κυρία Βασιλείου. Θέλω να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, γιατί δεν πρόκειται βέβαια μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ προσεκτικά δαπανούν τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Αυτό που που εγώ πιστεύω και ποια είναι η δικιά μου δέσμευση θα σας πω, ότι τα χρήματα πρέπει να δαπανώνται εκεί όπου άμεσα επηρεάζουν τους ανθρώπους και μπορούν να κάνουν μια διαφορά στον κάθε πολίτη της Ευρώπης ο οποίο από εμά προσδοκά να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε τη ζωή του. Ο πολιτισμό αποτελεί μέρο τη Ευρώπη, είναι μια βάση για την Ευρώπη και τα χρήματά μα πρέπει να τα δαπανάμε και στον πολιτισμό. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο τρόπο με τον οποίο δαπανάμε τα χρήματά μα είναι ο καλύτερο προκειμένου να βελτιώσουμε τη ζωή των νέων και γενικότερα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και ξεκινάω εγώ. Κυρία Βασιλείου, αναφερθήκατε στην εκπαίδευση των διδασκόντων και ρώτησε ήδη και ένα συνάδελφο κάτι σχετικό. Είστε διατεθειμένοι στο νέο πρόγραμμα διαβίου μάθησης να συμπεριλάβετε αυτό το θέμα και κυρίως όχι μόνο την περαιτέρω εκπαίδευση και τη βασική εκπαίδευση, αλλά την κινητικότητα οι δάσκαλοι οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ στο εξωτερικό δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν σωστούς Ευρωπαίους. Νομίζω πως ε, η Κομισιόν εδώ πέρα θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον ε, τομέα αυτόν. Παρακαλώ κύριε Βασίλη. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι πως ε, η κινητικότητα θα πρέπει να είναι δομημένη κινητικότητα, να μην έχει σκοπό τον τουρισμό. Να εξυπηρετεί ένα στόχο. Και οι μελέτες έχουν δείξει πώς η κινητικότητα βοηθάει όσους συμμετέχουν στο να αυξήσουν τις ε, δεξιότητές τους και τις ε, πιθανότητές τους για μια καλύτερη ζωή. Οπότε η κινητικότητα θα είναι τμήμα της ε, πολιτικής μας, αλλά όπως σας είπα μετά από προσεκτική μελέτη για να δούμε πού βρίσκονται τα εμπόδια στην κινητικότητα, ποια είναι τα ωφέλη και αφού διδαχτούμε και από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Αλλά η κινητικότητα θα παραμείνει ουσιαστικό τμήμα της ε, πολιτικής μας. Τώρα, για το ερώτημά σας για τους δασκάλους. Ναι, βεβαίως, πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να, έχουν, να επιδείξουν περισσότερη κινητικότητα. Ξέρω πως όταν κάποιος ε, ξεκινάει να δουλεύει δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να αφήσει πίσω την οικογένεια και να πάει στο εξωτερικό για να αποκτήσει εμπειρία, αλλά πρέπει να τους ενθαρρύνουμε. Να τους δώσουμε κίνητρα, γιατί η κινητικότητα των διδασκόντων είναι εξίσου σημαντική με την κινητικότητα των μαθητών και των λοιπόν βεβαίως. Λοιπόν, θα επανελθώ μια συμπληρωματική ερώτηση. Μπορείτε να μου υποσχεθείτε κυρία Βασιλείου, πως το νέο πρόγραμμα διαβίου μάθησης θα έχει ένα κομμάτι το οποίο θα λέγεται Comenius Teacher ή κάπως έτσι. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική μια τέτοια προσθήκη στο πρόγραμμα Comenius και σας είμαι ευγνώμων κυρία Πακ που προτείνετε μια τέτοια πτυχή για τους δασκάλους στο πρόγραμμα κομμένιους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά βεβαίως, ε, εφόσον πρόκειται για νέα πτυχή, πρέπει να την ενισχύσουμε για να αναπτυχθεί. Όπως ακριβώς και η, την ατομική κινητικότητα των μαθητών του κομμένιου, στην οποία ξεκινάμε φέτος, αλλά με 13 μόνο κράτη-μέλη. Γιατί? Γιατί δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένα ή δεν είναι πολύ σίγουροι για την ασφάλεια των νέων. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια, δηλαδή ότι το πρόγραμμα αυτό ε, ατομικής κινητικότητας θα διασφαλίζει την προστασία των 15χρονων ε, και 16χρονων που θα πάνε στο εξωτερικό με αυτό το πρόγραμμα. Οπότε ελπίζω φέτος. Σας ευχαριστώ κυρία Μπαντία. Ευχαριστώ, κυρία Βασιλείου. Έχετε και το χαρτοφυλάκιο για την πολυγλωσία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι από αυτού. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει το 2014 κάποιες αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη και το κριτήριο του πληθυσμού, πέρα από το κριτήριο το πόσες χώρες είναι. Η χρήση των γλωσσών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι έχουμε έναν ε, κανονισμό που από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία τη επιτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε πέντε χώρε στην αρχή με τρει μόνο γλώσσε. Σήμερα έχουμε 27 χώρε, 23 γλώσσε. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε κάποιε δυσκολίε όσον αφορά τη χρήση τη γλώσσα. Εσεί πώ βλέπετε τα πράγματα, θα μπορούσατε να σκεφτείτε να εξετάσετε τη δυνατότητα εισαγωγή του κριτηρίου και του πληθυσμού στον κανονισμό χρήσης των γλωσσών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Βασιλείου. Όπως ξέρετε, η χρήση των γλωσσών στηρίζεται σε κανονισμό του Συμβουλίου του 58. Και ο κανονισμός αυτός έχει τροπολογηθεί αρκετές φορές μετά από κάθε διεύρυνση και η τελευταία ήταν το 2007. Ο κανονισμός αυτός λέει ότι και οι 23 επίσημες γλώσσες θα πρέπει να είναι ίσες, να αναγνωρίζονται και να την χάνουν σεβασμού. Αλλά θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα. Διότι η συνθήκη μιλάει για ε, γλωσσική πολυμορφία και πρέπει να τη σεβόμαστε. Και η γλωσσική πολυμορφία δεν σημαίνει μόνο 23 γλώσσες. Σημαίνει περιφερειακές και μειονωτικές γλώσσες και έχουμε περίπου 60 τέτοιες. Και έχουμε άλλες 400 περίπου γλώσσες που μιλάνε οι μετανάστες στις κοινότητές τους. Πρέπει να κάνουμε πάσα δυνατή προσπάθεια να διατηρηθεί αυτή η ποικιλομορφία και να τη χάνει σεβασμού, γιατί είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής κουλτούρας και πολιτισμού αυτή η πολυμορφία και πρέπει να τη σεβόμαστε. Αλλά οποιαδήποτε τροπολογία του, του κανονισμού του Συμβουλίου είναι απόφαση του Συμβουλίου που πρέπει να λαμβάνεται αμόφωνα και δυστυχώς η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να κάνει προτάσεις στο Συμβούλιο για κάτι τέτοιο. Η κυρία Μπαντιά. Ναι, το γνωρίζω κυρία Βασιλείου. Αλλά βλέπετε, μετά από τόσα χρόνια που κατά τη γνώμη μου η χρήση της γλώσσας εδώ έχει δημιουργήσει κάποιες ανομαλίες, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ξανασκεφτούμε λίγο τα πράγματα. Ξέρω ότι είναι θέμα του Συμβουλίου, το γνωρίζω. Και ξέρω ότι δεν είναι και πολύ διατεθειμένοι να αλλάξουν τα πράγματα, όμως θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή εσείς να σκεφτείτε αυτό που σας λέω, ότι δηλαδή έχει νόημα για να στηρίξουμε την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη. Η κύριε Βασιλείου. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πιστεύω πάρα πολύ στην πολιτιστική πολυμορφία, ιδιαίτερα επειδή προέρχομαι από ένα μικρό κράτος νησιωτικό, κράτος νησί, και σας διαβεβαιώνω ότι με τα προγράμματά μας η πολιτική μας θα είναι να ενθαρρύνουμε την πολυγλωσία και την, πολιτική, την πολιτιστική πολυμορφία, ιδιαίτερα τη γλωσσική. Ό,τι είναι της αρμοδιότητάς μου και της αρμοδιότητας της, Κομισιο... της Επιτροπής θα το κάνουμε. Διότι πιστεύουμε σε αυτή τη γλωσσική ποικιλομορφία των λαών μας. Ο Σμιτ. Ευχαριστώ. Κυρία υποψήφια επίτροπε, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στα ουγγρικά για την ποικιλομορφία, μία από τις σημαντικότερες αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται και στις συνθήκες και ισχύει ιδιαίτερα και για τις μειονότητες που υπάρχουν στις ε, πατρίδες μας ε, οι λεγόμενες ε, αυτόφωνες μειονότητες οι οποίες θέλουν να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα τους στην διοίκηση. Στη Σλοβακία πρόσφατα πέρασε ένας νέος γλωσσικός νόμος που μεταχειρίζεται με διακριτικό τρόπο κάποιους ουγγρόφωνους πολίτες. Αναφέρω επιλέξει η σλοβακική γλώσσα έχει προφάδισμα έναντι όλων των υπολείπων και υπάρχει μάλιστα και πρόστιμο 5.000 ευρώ εάν χρησιμοποιήσει κανείς σε ε, συναλλαγές με το κράτος την ε, ουγγρική γλώσσα. Το γνωρίζω αυτό το νέο σλοβακικό νόμο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με πολύ προσοχή πώς εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Διότι εμείς ως Επιτροπή μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνο μέσω της εφαρμογής του τρόπου αυτού, του νόμου αυτού. Πώς εφαρμόζεται δηλαδή, και όπως πολύ καλά ξέρετε, η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο στην περίπτωση μειωνοτικών γλωσσών σε ορισμένες χώρες και γλωσσική πολιτική μόνο μέσω του Ευρω... της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν μπορούμε γενικά να παρεμβαίνουμε σε αποφάσεις κρατών μελών όσον αφορά γλωσσική πολιτική. Φυσικά τονίζω το ότι η προστασία των μειονοτήτων και των γλωσσών τους είναι τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει επικυρωθεί από όλε τι χώρε μέλη και οι χώρε μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν τι υποχρεώσει του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλε διεθνεί υποχρεώσει που έχουν. Αλλά η, η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτε παραπάνω από αυτού. Δέστε την κοινή δήλωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας και τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας που λένε ότι θα συνεργαστούν προκειμένου τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων να την χάνουν πλήρους σεβασμού. Επίσης συμφώνησα νομίζω ότι ο εκπρόσωπος θα τους συμβουλεύει στη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να εφαρμοστεί σωστά. Πάντως η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να φροντίσουμε να μην γίνει τίποτε το οποίο να είναι σε βάρος ή παράβαση της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Δευτερολογία. Η απάντησή σας με καθυσίχασε. Προφανώς γνωρίζετε την κατάσταση. Παρόλα αυτά φοβόμαστε γιατί καταργήθηκε η θέση της ε, πολυγλωσσίας ε, και συγχωνεύτηκε με το δικό σας ε, χαρτοφυλάκιο και επειδή και εσείς προέρχεστε από μια μικρή χώρα νομίζω πως και για εσάς θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να προστατεύσετε δηλαδή τις μικρές και μειονοτικές γλώσσες και έχετε γράψει στις γραπτές σας απαντήσεις πως θα κάνετε συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια είναι αυτά τα βήματα. Το ζήτημα των γλωσσών και της ε, πολυγλωσσίας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προσπαθήσουμε όχι μόνο να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την πολυγλωσσία, αλλά και να ενισχύσουμε τα προγράμματά μας για την ε, πολυγλωσσία. Και νομίζω πως ε, μέχρι το 2012 θα έχει εισαχθεί ένα νέο με ένας νέος δείκτης για την μάθηση ξαναγλωσσών από τους νέους, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την απόφαση 1 συν 2 και το πώς αυτή εφαρμόστηκε. Αλλά πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε κάθε παιδί να αρχίσει να μαθαίνει γλώσσες από μικρό. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Βασιλείου. Το πρόγραμμα Ζαμονέ είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διευκολυνθεί η γνώση όσον αφορά τη συνεργασία μέσα στην Ευρώπη. Ενισχύει την εκπαίδευση και τη σκέψη γενικά γύρω από την Ευρώπη. Το πρόγραμμα για την διαβίου μάθηση μέχρι το 2010 βοήθησε το πρόγραμμα Ζαμονέ και το Έρασμος και το Λονάρτο Νταβίντσι. Εν ώψη λοιπόν της προετοιμασίας του νέου προγράμματος διαβίου μάθησης, θέλω να ξέρω ποιες είναι οι δικές σας οι απόψεις για το πρόγραμμα Ζαμονέ και κατά πόσο θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να ενισχύεται. Ευχαριστώ. Το νέο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Ιδίως μάλιστα τα προγράμματα που έχουν στεφθεί με επιτυχία. Στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε από τη μέση προγράμματα επιτυχή, αλλά να τα ενισχύσουμε. Αν κάπου υπάρχουν αδυναμίες, να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Το Ζάμονε πράγματι ήταν ένα ιδιαίτερα επιτυχές πρόγραμμα, διότι συνδέει τους καθηγητές των πανεπιστημίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε έτσι να αποφεληθούμε από τη γνώση τους, από το ενδιαφέρον τους και επίσης είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος ώστε οι άνθρωποι στα κράτη-μέλη μας να μάθουν περισσότερα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, για το πώς δουλεύουμε εδώ, τι γίνεται εδώ. Το γεγονός επίσης ότι στηρίζουμε διάφορα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα που έχουμε επιλέξει, που αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτήν την ε, ιδέα την ευρωπαϊκή είναι πράγματα τα οποία θα συνεχιστούν. Στόχος μας πάντως δεν είναι να απαλείψουμε προγράμματα, αλλά να τα ενισχύσουμε. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Φίσα. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το νέο στάδιο με το χαρτοφυλάκιό σας έχετε και τις δράσεις Marie Curie, που μέχρι τώρα τις είχε Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα. Το σύστημα επιλογής των προγραμμάτων για αυτή τη δράση δείχνουν την ποιότητα και αυτό το λένε και όσοι έχουν ε, συμμετάσχει. Θα συνεχίσει το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα και που έχει οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα ή σκοπεύετε να το αλλάξετε. Η κυρία Βασιλείου. Πιστεύω πως ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος Μπαρός αποφάσισε τις δράσεις Μαρή Κιουρί να τις περάσει στη δικιά μου γενική διεύθυνση είναι επειδή ακριβώς θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το τρίγωνο της μάθησης εκπαίδευση, έρευνα και οι δράσει Marie Curie είναι ένα πάρα πολύ καλό ερευνητικό πρόγραμμα. Πρέπει όμως αυτά τα τρία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε από το μηδέν και δεν θα αναγνωρίσουμε την καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Καφέ άλλο. Εγώ σκοπεύω να συνεργαστώ στενά με τον αρμόδιο επίτροπο για την έρευνα προκειμένου να προχωρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τους ερευνητές και να τους ενθαρρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο όπως έγινε και κατά το παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα για να πλήξουμε το πρόγραμμα αυτό. Κάθε άλλο, μόνο για να εμπλουτίσουμε το τρίγωνο στο οποίο αναφέρθηκα και πριν. Ευχαριστούμε κυρία Νεβεντάλοβα. Ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την πολιτική όσον αφορά τους νέους και την διαδικασία λήψης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκείνοι δεν συμμετέχουν. Πιστεύουν οι νέοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται για την νεολαία. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς προβλέπετε κάποιο πλαίσιο που να έχει να κάνει για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών και πώς θα προχωρήσει αυτό στη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Επίσης για το σύμφωνο για την Ευρωπαϊκή Νεολαία. Ε, άκουσα τη μία σας ερώτηση για την ε, αδιαφορία που νιώθουν οι νέοι από πλευράς της Ευρώπης προς το μέρος τους και για την απόσταση αυτή ανάμεσα στον κόσμο τους νέους κυρίως και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει πάρα πολλές κοινωνίες στα κράτη-μέλη. Πρέπει να προσελκύσουμε τον ενδιαφέρον των νέων. Και αυτό είναι μια προσθήκη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει όμως να αναλάβουμε δράση, ώστε να κάνουμε τον κόσμο να ενδιαφερθεί περισσότερο στη δημοκρατική ζωή των κοινωνιών. Αυτό αποτελεί ένα κεντρικό σημείο των προγραμμάτων μας για το μέλλον. Το πώς δηλαδή θα κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των νέων μας, ώστε να ενδιαφερθούν περισσότερο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά και τα περιφερειακά και τα τοπικά και τα εθνικά. Είναι μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης ε, του στήματος του συμμετέχει. Πώς να νιώθουν οι άνθρωποι ότι η Ευρώπη τους ανήκει και ότι αποτελούν μέρος της. Είναι μέρος της ε, πολιτικής μας. Και όχι μόνο της Ευρώπης και των εθνικών χωρών πρέπει να είναι, των κρατών. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό που ρώτησα είναι το εξής. Τι πιστεύετε για αυτά τα θέματα συγκεκριμένα. Χαίρομαι που λέτε ότι πρέπει να τους δώσουμε περισσότερη σημασία. Ναι, αλλά τι θα κάνετε για να το πετύχετε αυτό. Και τι πιστεύετε για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 σε σχέση πάντα με την νεολαία και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την νεολαία. Η κυρία Βασιλείου. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Έχουμε ειδικά τμήματα στα προγράμματά μας που απευθύνονται ακριβώς αυτό το στόχο, δηλαδή συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Θα τα ενισχύσουμε τα προγράμματα αυτά, θα τα εμπλουτίσουμε, γιατί όπως είπα και πριν, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των νέων για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στις χώρες τους, στους δήμους τους, στις περιοχές τους, είναι κάτι πολύ σημαντικό. το διαπιστώσαμε ότι υπάρχει απόσταση με τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτή η αδιαφορία των νέων. Για τη στρατηγική 2020, βεβαίως, οι νέοι αποτελούν μέρος της όλης πολιτικής μας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, νέες δεξιοτεχνίες. Μα οι νέοι είναι το μέλλον μας. Αν δεν φροντίσουμε για τους νέους, για ποιους θα φροντίσουμε. Είναι το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λόκεκαρτ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζώντας οικονομική ύφεση, όπως σωστά είπατε κι εσείς, ακόμα και οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων δεν βρίσκουν δουλειά και οι επιχειρήσεις υφίστανται όντω και πια τον ανταγωνισμό παγκόσμια. Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το διάλογο μεταξύ τη βιομηχανία και του εκπαιδευτικού κόσμου. Α το πούμε γι' αυτό τα σχολεία, τα πανεπιστήμια πρέπει να εξυγχρονιστούν, πρέπει να υπάρχουν στρατηγικέ συμφωνίε μεταξύ τη βιομηχανία και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να δώσουν νέε ευκαιρίε μεταφορά των γνώσεων και νέου τρόπου χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Υποθέτοντας ότι η υποψήφια συμφωνεί με αυτόν τον προβληματισμό και το πιστεύω αυτό, ερωτώ Πώς σκοπεύετε περαιτέρω να ενισχύσετε αυτή τη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνολογίας αμφίδρο μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων. Απάντηση. Νομίζω ότι αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας υπήρξε επιτυχής μέχρι σήμερα. Βλέπουμε τα ωφέλη. Πριν αναφέρθηκα στο πώς μπορούμε να συνδέσουμε τις δεξιότητες με την απασχόληση να έχουν τη δυνατότητα όλοι να βρούνε δουλειά αλλά αν στηριχτούμε στις καλές εμπειρίες που είχαμε με το φόρουμ αυτό Πανεπιστημίων Βιομηχανίας θα πρέπει να το επεκτείνουμε σε επαγγελματική κατάρτιση αυτό είναι σημαντικό προγράμματα για το να μπορούν να πηγαίνουν οι φοιτητές σε βιομηχανίες γιατί είναι χρήσιμο, τους δίνει πρακτική εμπειρία, όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις και, και θα πρέπει να το επεκτείνουμε και στα, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με τη βιομηχανία. Έχω εμπειρία από την Κύπρο όπου μία εβδομάδα κάθε χρόνο κάθε απόφυτος ενό σχολείο θα πρέπει να πάει δίπλα σε κάποιον που ασκεί ένα επάγγελμα να πάρει την εμπειρία, να δει την εμπειρία πρακτικά. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή τοποθέτηση σε θέσεις στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχετε δίκιο λοιπόν. Αυτό το φόρουμ βιομηχανία πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και θα πρέπει να επεκταθεί και στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Δευτερολογία μου θα είμαι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχουμε πετυχημένα εργαλεία, όπω είπατε, για την εταιρική αυτή σχέση στα κράτη-μέλη, στη Δανία, τη χώρα μου, έχουμε το λεγόμενο βιομηχανικό PhD. Έχουμε πανεπιστήμια, μία επιχείρηση και το κράτο. Τρίγωνο. Έπειτα ένας ε, απασχολούμενο σε μια επιχείρηση μπορεί να πάρει ένα PhD που τη δίνει το πανεπιστήμιο και το κράτος ε, ή δέχεται ή απορρίπτει το αίτημα της επιχείρησης. Αν εγκριθεί, παίρνει μια επιδότηση από το κράτος η επιχείρηση. Ο υπάγγελο μοιράζει το χρόνο του 50-50 μεταξύ της επιχειρησης αν εγκριθει παιρνει μια επιδοτηση απο το κρατος η επιχειρηση ο υπάλληλο μοιραζει το χρονο του 50 50 μεταξυ της επιχειρησης και του πανεπιστήμιου. Εσείς ως επίτροπος σκοπεύετε να εισάγετε αυτό το βιομηχανικό PhD όπως γίνεται στη Δανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρξουν και, τα, και να φροντίσετε να υπάρξουν τα αναγκαία κονδύλια απάντηση. Πρέπει να το μελετήσω αυτό που λέτε προσεκτικά, να δω πώς λειτουργεί και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα και είμαι σίγουρη επειδή η δουλειά μας στηρίζεται στη συνεργασία και ανταλλαγή των άριστων μεθόδων αν πιστούμε ότι αυτό το δανέζικο παράδειγμα είναι μια καλή πρακτική η πολιτική μου θα είναι καλή πρακτική σημαίνει καλή πολιτική. Αν λοιπόν πιστούμε ότι είναι μια καλή μέθοδος, με το διάλογο που θα έχουμε, μπορεί να το εγκρίνουμε ως δική μας καλή πολιτική. Η κυρία Σάντσες Σμιτ, κυρία Βασιλείου, στην αρχή αναφερθήκατε στην ενότητα μέσα στη διαφορά. Μιλήστε για τη συνθήκη, για την πρόθεση της πικρομορφίας των πολιτισμικών εκδηλώσεων UNESCO. Η συνθήκη τη Λισαβόνα, αν δεν μέσα στου στόχου τη έχει την αναφορά σε αυτό το σεβασμό τη πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία. Τι μέτρα θα λάβατε προκειμένου να ευνοήσετε την πολιτισμική ε, ποικιλομορφία και στο ιστορικό τη Ένωση και στις σχέσεις με τις λιγότερα αναπτυγμένες χώρες, πολιτική γειτονία, Μεσόγειο κλπ. Η κυρία Βασιλείου θα απαντήσει. Ένας από τους στόχους μας είναι να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την πολιτισμική ποικιλομορφία και την επικύρωση της συνθήκης της UNESCO. Διάβασα με μου ότι δύο χώρες μέλη ακόμα δεν το έχουν επικυρώσει. Δεν λέω ποιες είναι. Ελπίζω σύντομα να επικυρώσουν και αυτές. Υπάρχει μια υποψήφια χώρα που δεν έχει ακόμα επικυρώσει. Ελπίζω και αυτή να το επικυρώσει. Και πρέπει να προωθήσουμε την πολιτισμική ποικιλομορφία στη σχέση μας με τον έξω κόσμο. Να προωθήσουμε την επικύρωση αυτής της συνθήκης εννοούμε παγκόσμια. Με ευχαρίστηση άκουσα, διάβασα μάλλον, στα πορίσματα της πρόσφατης διάσκεψης κορυφής Ένωση Κίνα, ένα από τα θέματα που ετέθησαν στο κοινό ανακοινωθέν είναι ότι η Ένωση και η Κίνα θα προωθήσουν την επικύρωση αυτής της συνθήκης. Προωθούμε την πολιτισμική ποικιλομορφία και με πολλές άλλες τρίτες χώρες, διότι ε, δεν ζούμε σε απομόνωση, ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο χώρο και η πολιτισμική ποικιλομορφία και ο σεβασμός της για όλους τους λαούς θα πρέπει να είναι μια από τις βάσεις για τη σχέση μας με τον έξω κόσμο. Και υπάρχουν πρωτόκολλα με πολλές χώρες για το θέμα αυτό. Τονίζω και υπογραμμίζω το ότι στις διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες υπάρχει προϋπόθεση ο, ήδη να έχουν επικυρώσει τη συνθήκη αυτή τη συνθήκη για την πολιτισμική ποικιλομορφία. Το θεωρούμε άκρος αναγκαία προϋπόθεση για μια τέτοια σχέση. Η Μαρή Τερέζ θα δευτερολογήσει. Για το πρωτόκολλο αυτό να εισαχθεί το πρωτόκολλο πολιτισμική συμφωνία στι εμπορικέ συμφωνίε με τι χώρε. Ποια είναι η γνώμη σα από αυτού. Απάντηση. Θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι στο πώς προωθούμε την πολιτισμική ποικιλομορφία. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι ένας καλός τρόπος πρόθεσης του πολιτισμού, γιατί όπως είπα και πριν, ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση πολιτισμικών διαφορών μεταξύ μας είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για οποιοδήποτε άλλη σχέση. Αν λοιπόν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες, θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι σίγουροι ότι τη χάνει σεβασμού η πολιτισμική ποικιλομορφία. Ευχαριστώ κύριο Σίβαν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα ερώτημα το οποίο μου το έστειλε το κοινό και θα σας το διαβάσω. Ετέθη ενισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και έχει νέες αρμοδιότητες στον τομέα του αθλητισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε για το μέλλον του αθλητισμού για να προωθήσετε τον αθλητισμό ως καταλήτη της κοινωνικής συνοχής, της ένταξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Κυρία Βασιλείου, όπως είπα και σε άλλη ερώτηση, ο αθλητισμός έχει μια ξεχωριστή πολύ σημαντική πτυχή. Είναι ο κοινωνικός ρόλος. Και σκοπεύω πραγματικά να δώσω βάρος εκεί πέρα. Γιατί βεβαίως ο αθλητισμός είναι αυταξία, αλλά είναι και μέσον για άλλες ε, πολιτικές. Π.χ. έχω την εμπειρία της υγείας σχετίζεται με τη σωματική δραστηριότητα. Και έχουμε μελέτες που δείχνουν σαφώς πως η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για παχυσαρκία και γενικότερη κακή υγεία. Τώρα, έχουμε και τα προγράμματα του 2009-2010 για να ανοίξουν το δρόμο για πιο μόνιμα προγράμματα στον τομέα του αθλητισμού. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτά, να δούμε πώς ε, θα εφαρμόσουμε τις νέες μας αρμοδιότητες ε, σύμφωνα με την συνθήκη. Βλέπω πως υπάρχουν πολύ σημαντικές πτυχές στον αθλητισμό εδώ πέρα, όπως η ισότητα, η κοινωνική πτυχή του αθλητισμού, η συνεισφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Τώρα πρέπει να δούμε ζητήματα όπως η βία, ο ρατσισμός, ε, Όλες αυτές ε, οι πτυχές είναι πάρα πολύ σημαντικές και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, στο να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση, όχι. Ναι. Ο κύριος Σβέρ. Κυρία Υποψήφια Επιτροπή, έχω ένα πιο γενικό ερώτημα. Θετικό είναι ότι αναφέρατε στην αρχή την ε, ένωση μέσα από την ε, ποικιλομορφία και πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια sui generis οντότητα. Υπάρχει η διαδικασία της Κοπενχάγης, η διαδικασία της Μπολόνιας, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα και αναφέρατε κάποια από αυτά. 80 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση και από την άλλη μόνο ένα δέκατο των Ευρωπαίων είναι στην διαβίου κατάρτιση. Πάρα πολλά παιδιά σταματάνε το σχολείο, δεν τελειώνουν το σχολείο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα. Θεωρείται πως η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού εξακολουθεί να αποτελεί την κατάλληλη βάση συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, νομίζω πως ναι. Στον τομέα αυτών νομίζω πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε να επιτελέσουμε το έργο μας. Το πρόβλημα είναι πως πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος στην εμπειρία. Όπως είπα πριν με κάποια άλλη ευκαιρία. Έχουμε διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές ιδέες στα κρατη Δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε. Απλά πρέπει να δεχτούμε από τις καλές πρακτικές των άλλων. Όχι να αντιγράψουμε, να δούμε πώς αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και να δούμε πώς μπορούμε μετά να προσαρμόσουμε αυτή την απάντηση στον εθνικό περιβάλλον. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος και αυτό αποδείχθηκε και με τη διαδικασία της Μπολόνια. Γνωρίζετε πως στην αρχή, ξέρω πως ε, οι υπουργοί ήταν πολύ επιφυλακτικοί και υπάρχουν ακόμα προβλήματα με τη διαδικασία της Μπολόνιας. Ε, δεν έχουμε 100% επιτυχία, αλλά σε μεγάλο βαθμό είχαμε επιτυχία και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την ε, συνεργασία και σε άλλους τομείς. Ε, αναφέρω εδώ πέρα παραδείγματο χάρη την ε, επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν πάρα πολύ στενά με τα κράτη-μέλη. Γνωρίζω παραδείγματο χάρη πως υπάρχουν πολύ καλά ΙΕΚ ε, στην Τσεχία. Να δούμε λοιπόν πως μπορούμε να τα εξυγχρονίσουμε και να αναγνωρίσουμε τα διπλώματα τα οποία δίνουν για να διευκολύνουμε ακριβώς την διάχυση της γνώσης ε, και της εμπειρίας. Ε, έχετε συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα δεν έχουν ε, πολλές δυνατότητες άμεσης παρέμβασης και διαμόρφωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη, αλλά μπορείτε να επιταχύνετε κάποιες διαδικασίες, π.χ. την πολυγλωσία στα σχολεία. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια η ιδέα ενός ευρωπαϊκού γλωσσικού δίκτυ ήταν πολύ επίκαιρη, είχε προωθηθεί από τον Επίτροπο Φίγκελ. Αργότερα δεν ξανακούσαμε για αυτή την ιδέα. Θέλω λοιπόν να ακούσω την άποψή σας. Έχετε καμία σοβαρή πρόθεση για την ε, έρευνα των γλωσσικών ικανοτήτων των νέων και να ξαναξεκινήσουν αυτές τις μελέτες. Η κυρία Βασιλείου. Ναι, πιστεύω πως ε, είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί το πιστεύω, εγώ έχω δύο κόρες παντρεμένες, έχω εγγόνια και πάντα λέω στις κόρες μου μετανιώνω το ότι εγώ όταν ήμουν νέα δεν είχα πολλές ευκαιρίες να μάθω γλώσσες. Προσπαθώ λοιπόν τώρα να μάθω γλώσσες και είμαι και υπεύθυνη πολυγλωσσίας. Πρέπει να κάνω περισσότερα. Αλλά είναι δύσκολο στην ηλικία μου. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τα μικρά παιδιά. Είναι φανταστικό το πώ τα παιδιά πόσο εύκολα μαθαίνουν. Ε, σας σφουγγάρια. ό,τι ακούνε το μαθαίνουν. Δεν νομίζω να μπερδεύονται. Έχω δει παιδιά από γάμους ε, δύο γονιών με διαφορετικές γλώσσες που μιλάνε τη γλώσσα του κάθε γονιού και μία τρίτη στο σχολείο. Οπότε τα παιδιά μπορούν να μάθουν και πρέπει να του δίνουμε την ευκαιρία να μάθουν περισσότερες γλώσσες. Όχι μόνο για να μάθουν, αλλά ως μέσο για μια καλύτερη ζωή. Ο κύριο Μπέλετ. Κύρια Βασιλείου, θα ήθελα να επανέλθω στον τομέα του αθλητισμού και συγκεκριμένα στην έλλειψη νομικής βεβαιότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές πώς πρέπει να δούμε την ε, διακυβέρνηση που γίνεται κατά περίπτωση. Αυτό ισχύει ειδικά σε τρία ζητήματα συλλογικές πωλήσει δικαιωμάτων ΜΜΕ, δημόσια χρηματοδότηση του αθλητισμού, των υποδομών και οι πράκτορες των παικτών. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά, ειδικά με τις νέες αρμοδιότητες Λισαβόνας. Υπάρχουν στον τομέα του αθλητισμού πολλές προσδοκίες και το ερώτημα μου είναι πολύ συγκεκριμένα. Σκοπεύετε να προετοιμάσετε κατευθυντήριες γραμμές για να υπάρχει περισσότερη νομική βεβαιότητα. Όπως σας είπα, συλλογικά δικαιώματα, πράκτορες παικτών κτλ. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορούμε να έχουμε γενικό, γενικούς κανόνες. Πρέπει αυτό να γίνει κατά περίπτωση. Και αναφέρατε τρεις περιπτώσεις και είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ με τις υπηρεσίες μου, αλλά κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό, με το αθλητικό κίνημα για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης πρέπει να συνεργαστώ με τους ε, υπόλοιπους επιτρόπους, γιατί υπάρχει εδώ πέρα ευρωπαϊκό δίκαιο που ισχύει του ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς, ε, της ελεύθερης ε, διακίνησης, ελεύθερης πρόσφορας υπηρεσιών, ζητήματα πολύ σημαντικά του ευρωπαϊκού δικαίου που πρέπει να γίνουν σεβαστά, αλλά πρέπει να δούμε πώς η ιδιαιτερότητα του αθλητισμού θα γίνει σεβαστή για να βρούμε την ε, καταλληλότερη λύση για να επιτύχουμε το στόχο που αναφέρατε. Ε, συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Μπέλετ. Ευχαριστώ, κύριε Πακ. Να επαναλάβω την ερώτησή μου για κατευθυντήριε γραμμέ. Είστε διατεθειμένοι να συντάξετε κατευθυντήριε γραμμέ. Και μετά, για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, κυρία Βασιλείου. Είναι άλλη μια πρόκληση και πιο συγκεκριμένα το γεγονός πως υπάρχει κάποια αντίφαση, αν θέλετε, με την ιδιωτική σφαίρα των αθλητών. Ποια είναι η άποψή σας ε, για τον κώδικα καταπολέμησης του ντόπινγκ της WADA, ε, ε, της Παγκόσμιας Υπηρεσίας που ασχολείται με αυτό το θέμα και αν σκοπεύετε να τον αλλάξετε. Για το πρώτο σας ερώτημα, να δούμε να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες μας, να δούμε τι λένε, αν οι κατευθυντήρες γραμμές μπορούν να μας βοηθήσουν. Θα το συζητήσω αυτό με την νομική υπηρεσία και με τους άλλους επιτρόπους που τους ενδιαφέρει το θέμα. Αν οι κατευθυντήρες γραμμές είναι λύση. Σας υπόσχομαι ωστόσο ότι είμαι διατεθειμένη να ακούσω με διάλογο οτιδήποτε. Σχετικά με το αντι-doping τώρα. Είχαμε ένα διάλογο με την ΟΑΤΑ. Η ΟΑΤΑ βελτίωσε τους, τους κανόνες της πάρα πολύ. Βέβαια, κι άλλη βελτίωση μπορεί να επέλθει. Πάντως, η προσωπική μου γνώμη και το συγκεκριμένο αυτό κανόνα είναι ότι πρέπει να εφαρμόζουμε τον κανόνα της αναλογικότητας. Είναι αυτό ανάλογο σε σχέση με το δικαίωμα του σεβασμού του ιδιωτικού χώρου. Έχουμε στο Βέλγιο ένα πρόσφατο παράδειγμα που αποκλείστηκαν πέντε παίχτες για έναν χρόνο επειδή δεν τηρήθηκε αυτός ο κανόνας του whereabout όπως το λέμε. Πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου από αυτό. Πάντως η Επιτροπή θα μελετήσει την περίπτωση διότι υπήρξε καταγγελία. κύριος Φλέκενστάιν. Κυρία Επίτροπε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ήδη ένα δίκτυο εθνικών πολιτισμικών Ινστιτούτων, το UNIC, που αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας αυτών των Ινστιτούτων για το πώς θα επιτελέσουν πολυπολιτισμικά έργα και πρωτοβουλίες. Πώς βρίσκεται την πρωτοβουλία των να αποτελέσουν αυτά κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Ε, Κυρία Βασιλείου, ναι, ανέφερα πριν ε, την σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική ποικιλομορφία και βεβαίως έχουμε ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε το πώς θα κυρωθεί ανά τον κόσμο, αλλά και να συμπεριλάβουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία στη σχέση μας με τον έξω κόσμο. Γιατί όπως είπα, ζούμε σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο, πρέπει να σεβαστούμε την πολιτιστική ποικιλομορφία και οι πολιτιστικές ανταλλαγές και σχέσεις μεταξύ Ένωσης και άλλων χωρών είναι πολύ σημαντικές ε, στο να αυξηθεί η άλλη αλληλοκατανόηση και στο να έρθουν πιο κοντά οι λαοί μας. Οπότε είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση κύριε Φλέκενστάιν. Ναι, θα είμαι σύντομος. Θα αναφερθώ στο τελευταίο κομμάτι της απάντησής σας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα οργανώσετε κάτι τέτοιο ή θεωρείτε πως είναι υπόθεση των κρατών μελών. Δηλαδή, πώς θα συμπεριλάβετε κάτι τέτοιο στην πολιτική σας. Παρακαλώ κύριε Βασιλείου. Ε, εξαρτάται τι εννοείτε να οργανώσω. Εάν εννοείτε να συνεργαστούν τρίτες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κάνουμε ήδη και ήδη έχουμε προγράμματα που ενθαρρύνουν τις ε, πολιτισμικές ε, ανταλλαγές, την προώθηση των ξένων πολιτισμών στην Ένωση και αντιστρόφως. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Διεθνούς ε, στη Σανγκάη σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση ως ένα μέσο προώθησης του πολιτισμού και της ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα και στους επισκέπτες από τις άλλες χώρες αλλά αυτό το έχουμε κάνει και με άλλες χώρες, στις Βρυξέλλες και σε πολλές άλλες χώρες είμαι σίγουρη. Χτες π.χ. μιλώντας με τις υπηρεσίες μου άκουσα πως όταν το Λίβερπουλ ήταν πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης είχαν μια έκθεση Ινδικής τέχνης, Κινέζικης τέχνης, Αφρικανικής τέχνης και αυτό είναι ένας τρόπος ε, να προωθηθούν αυτές οι ανταλλαγές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βάτιμο. Ευχαριστώ πολύ. Έδωσα μία ερώτηση στα γαλλικά, μπορείτε να τη διαβάσετε, αλλά θα τη συνοψίσω. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στις χώρες μας έχουν συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κάθε χώρα στο πώς προωθείται η εργασία των φοιτητών, η βοήθεια, οι υποτροφίες, φοιτητικές αιστείες. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Ιταλία που έχουν 300.000 εγγεγραμμένους φοιτητές. Και ρωτώ μπορεί η Ευρώπη να κάνει κάτι έτσι ώστε η κάθε χώρα να προωθήσει καλύτερα όλες αυτές τις επιπλέον πτυχές παράλληλα που είναι αναγκαίες για την πανεπιστημιακή κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων, η κυρία Βασιλείου. Ξέρω ότι υπάρχει, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το που κάνουν για την κινητικότητα των φοιτητών, για τις υποτροφίες, τη στέγασή τους, τις μεταφορές, συγκοινωνίες ενώ κλπ. Μεγάλη διαφορά. Ξέρετε όμως τους περιορισμούς μας. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη, στα πανεπιστήμια γιατί ένας από τους στόχους μας είναι να έχουμε αυτόνομα, ανεξάρτητα πανεπιστήμια. Άρα πρέπει να σεβόμαστε την αυτονομία τους. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε, να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να το κάνουν, διότι αν δουν την χρησιμότητα και το ενδιαφέρον των φοιτητών τους από την κινητικότητα προς το εξωτερικό, θα το κάνουν και για τους ξένους φοιτητές στη χώρα τους. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που δίνει ε, χαμηλό το καδάνια σε φοιτητέ. Αυτό εξαρτάται όμως από διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της κάθε χώρας και της τράπεζας. Εμείς ενθαρρύνουμε την τράπεζα να έχει ένα ενιαίο σύστημα για φοιτητικά δάνεια για κάθε χώρα. Φυσικά η κάθε χώρα θα πρέπει να συμφωνήσει ποιος θα διαχειρίζεται αυτά τα δάνεια. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος ενθάρρυνσης της κινητικότητας των φοιτητών. Δευτερολογία του κυρίου Βάτιμο. Εγώ και εγώ έχω απάντηση. Είχα κατά νου ένα κριτήριο Μάστριχτ για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων ευρωπαϊκά. Δηλαδή, αν σε μια χώρα τα πανεπιστήμια δεν πετύχουν ένα αλφα ποσοστό υποτροφιών ή αν παρά είναι μεγάλα, τους μειώνεται η δυνατότητα να αναγνωρίζετε το πτυχίο τους. Ένα είδος επιβολής εκ μέρους της Ένωσης θα μπορούσε να γίνει πιέζοντας μέσω της διεθνούς αναγνώρισης των τίτλων σπουδών. Απάντηση. Σας υπόσχομαι ότι τον επόμενο Μάρτιο που δέχουμε την Υπουργική Διάσκεψη για την διαδικασία της Μπολόνια δέκα χρόνια ζωής της διαδικασίας αυτής και θα συνιστούν οι Υπουργοί στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι θα το συζητήσω με του υπουργού. Γιατί βλέπω τα ωφέλη. Αλλά οι υπουργοί θα πρέπει να αναλάβουν την κίνηση. Πρέπει και αυτοί να δούνε τα ωφέλη. Πρέπει και αυτοί να δούνε τι δυνατότητες έχουν. Γιατί αυτό συνεπάγεται δημοσιονομικέ επιπτώσεις. Αν κάθε χώρα κάθε χώρα έχει διαφορετική κατάσταση. Θα το συζητήσω με τους υπουργού να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Πρόεδρος. Κύριος Βάτη μου ευχαριστεί. Πρόεδρος. Κυρία Βασιλείου. Κυρία Βασιλείου, συγγνώμη που μιλάω πίσω σας. Η κυρία Τρίπελ, τονίσατε την ανάγκη να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ αφενός, αφετέρου σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Σήμερα που ξέρουμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε ένα πολιτικά κατευθυνόμενο, ελεγχόμενο ίντερνετ όπως στην Κίνα και στην Ιράν, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να βρούμε καλά μοντέλα και λύσεις για αυτή την ισορροπία. Θα ήθελα τη γνώμη σας από αυτό. η κυρία Βασιλείου. Αδιαμφισβήτητα, κανένας δεν αφιβάλλει δηλαδή, ότι με τις εξελίξεις της τεχνολογίας πρέπει να παραμείνουν τα δικαιώματα του δημιουργού, τα πνευματικά δικαιώματα. Σωστά αμοιβόμενα για το έργο τους. Διαφορετικά δεν θα έχουμε δημιουργικό έργο. Χρειάζεται ανταμοιβή, αλλά όπως είπατε Ταυτόχρονα πρέπει οι νέες τεχνολογίες αυτές να ανοίξουν σε καλύτερη πρόσβαση για τους πολίτες μας, για γνώσεις και πολιτισμό. Υπάρχουν ακαθόδη θέματα εδώ. Αυτό που σας υπόσχομαι είναι ότι θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους επιτρόπους για τον ανταγωνισμό, τον Επίτροπο, τον Επίτροπο της Εσωτερικής Αγοράς για το πώς θα βρεθεί η πιο καλή λύση και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα και άλλα συναφή, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, πώς μπορούμε να τις συνδυάσουμε αφενός τα συμφέροντα των συγγραφέων και των εκδοτών και απ' την άλλη τα συμφέροντα των αναγνωστών και του κοινού που θέλουν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε βιβλία και λογοτεχνικά έργα. Πρέπει να πετύχουμε μια λεπτή ισορροπία. Και αυτό απαιτεί ειλικρίνεια και διάλογο μεταξύ των επιτρόπων και μεταξύ όλων των πρωταγωνιστών και ενδιαφερομένων σε αυτό. Η κυρία Τρίπελ δευτερολογία. Δηλαδή, σκοπεύεται να γίνουν κοινέ διασκέψει με του διάφορου ενδιαφερόμενου και με του συναδέλφου επιτρόπου για να πετύχετε μια ρεαλιστική, ισορροπημένη λύση. Απάντηση. Φυσικά. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Ξέρω ότι υπήρξαν ορισμένε πρωτοβουλίε στο παρελθόν. Τώρα χρειάζεται συντονισμός η Επιτροπή πρέπει να συντονίσει σε στενή συνεργασία, όπως είπα, με όλους τους σημαντικούς ενδιαφερόμενους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το συμφέρον όλων των πλευρών. Ο κύριος Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πακ. Ευχαριστώ και την κυρία Βασιλείου που ήρθε εδώ. Υπάρχουν ε, δύο μόνο προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που στοχεύουν τους νέους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά από τον χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής ε, και αναφέρομαι μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα Erasmus Mundus το οποίο αναφέρατε. Πώς θα βλέπατε την δυνατότητα αύξησης των κονδυλίων για αυτά τα προγράμματα. Στο πρόγραμμα δε το οποίο εσείς προτείνατε το νεολαία σε κίνηση. Το πρόγραμμα αυτό θα στοχεύει και στους νέους της λεγόμενης ανατολικής γειτονίας. Ναι, ελπίζω ναι. Ελπίζω να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και αυτούς τους νέους, αλλά πέρα από το Erasmus Mundus, ε, το οποίο νομίζω είναι φανταστικό πρόγραμμα και πρέπει να το ενισχύσουμε και να το δώσουμε νέα ορμή, να μην ξεχνάμε τη νέα προσθήκη που έχουμε, το Marie Curie, που είναι φανταστική ευκαιρία για τους νέους ερευνητές, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός, να συνεργαστούν με τους δικούς μας έρευνητές και να εμπλουτίσουν έτσι τις εμπειρίες που έχουν στον τομέα έρευνας τους. Από την δική μου πλευρά και είναι κατανοητό για να δοθεί ορμή σε όλα αυτά τα προγράμματα βεβαίως θα προσπαθήσω να αποκτήσω μεγαλύτερο προϋπολογισμό αλλά εδώ θα χρειαστώ την βοήθειά σας. γιατί τώρα βεβαίως ξεκινάνε οι νέοι οι νέες διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορώ εγώ τώρα να δεσμευτώ, αλλά θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ο πολιτισμός, η πολυγλωσία, η εκπαίδευση να ληφθούν υπόψη στο νέο πλαίσιο. Κύριε Μιγκάλσκι. Θα μπορούμε νομίζω να σας διαβεβαιώσουμε κύριε Βασιλείου για την στήριξή μας και θα ήθελα να ζητήσω και την δική σας διαβεβαίωση, μια δέσμευση πως όχι μόνο θα κάνετε ό,τι μπορείτε και θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια, θα ήθελα μια διαβεβαίωση ότι τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα για τα υπάρχοντα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους από την Ανατολική Ευρώπη που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχυθούν αυτά τα συγκεκριμένα κονδύλια. Και θα ήθελα μια διαβεβαίωση πως θα υπάρχουν αρκετοί πόροι έτσι ώστε αυτοί οι νέοι να χρησιμοποιήσουν την δική μας εμπειρία. Η κυρία Βασιλείου, ευχαρίστως πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας δώσω μια τέτοια διαβεβαίωση. Μακάρι να μπορούσα να σας το εγγυηθώ, αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Είναι σαν, να ζητάτε από έναν υπουργό στην χώρα σας, ε, τον Υπουργό Παιδείας, να σας πει το, εάν θέλει αυξημένο προϋπολογισμό. Ε, οπωσδήποτε. Αυτός ή αυτή θέλει παραπάνω προπολογισμό, οπότε και εγώ το ίδιο. Αλλά χαίρομαι που ακούω πως θα έχω τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Ε, δεν έχω αμφιβολία γιατί ξέρω πόσο πολύ είναι ε, στο πλευρό μας τα, μέρη, τα μέλη αυτής της Επιτροπής αλλά θέλουμε βεβαίως και τη στήριξη των κρατών μελών, του Συμβουλίου δηλαδή, των ενδιαφερομένων γιατί ο ρόλος τους, η πίεση δηλαδή που θα ασκήσουν για να ζήσουν περισσότερα κονδύλια δηλαδή, παίζει σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ κύριε Μπίσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην στρατηγική της νεολαίας γίνεται λόγος για ψηφιακή ένταξη, ψηφιακή συμπερίληψη και έχω ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Αν έχετε κάποια ιδέα ήδη για το ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε έτσι ώστε να προωθηθεί η ψηφιακή ένταξη των νέων. Παρακαλώ κυρία Βασιλείου. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη που υπάρχει προκειμένου νέες τεχνολογίες να συμπεριληφθούν στη δουλειά μας. Χρειάζεται κατάρτιση και παντού χρειάζεται, ακόμα και στον πολιτισμό χρειάζεται να ξέρουμε τα ψηφιακά μέσα. Υπάρχει το νέο πρόγραμμα Media. Τον επόμενο χρόνο περνάει στη ψηφιακή μορφή. Εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να το στηρίξουμε. Αλλιώς καταλαβαίνετε ότι θα μείνουμε απ' έξω. Θα έχουμε μόνο μερικούς μεγάλους κινηματογράφους που θα βάζουν τα μεγάλα ε, αμερικανικά, βραζιλιάνικα, δεν ξέρω εγώ τι έργα. Δεν λέω ότι έχω κάτι εναντίον τους, αλλά θέλω και ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας να προωθηθεί. Πρέπει όμως να περάσει σε ψηφιακή μορφή. Άρα το ψηφιακό έργο είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Και αυτό ακριβώς έχουμε συμπεραλάβει στη νέα μας στρατηγική. Συμπληρωματική. Α, όχι. Ο κύριος Σκέλη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πολύ που σας άκουσα να μιλάτε με ενθουσιασμό για τον αθλητισμό που είπατε πόσα θετικά κάνει για τον ε, πληθυσμό. Μας είπατε ότι το τελευταίο τμήμα της παρουσίασής σας ε, ήταν για τον αθλητισμό αλλά δεν προλάβατε να μας το παρουσιάσετε. Μπορείτε να μας το δώσετε παρακαλώ. Έπειτα, στον κατάλογο των προτεραιοτήτων σας, από τις γραπτές απαντήσεις σας, τον αθλητισμό το βλέπουμε μόνο δύο φορές στις γραπτές απαντήσεις σας. Κάπου που μιλάτε για τη Λισαβόνα και που λέτε ότι ελπίστε το 2011 να μπορέσετε να κάνετε προτάσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Άμα είναι τόσο σημαντικό ο αθλητισμός, γιατί να μην ξεκινήσουμε από το 2010 αλλά να περιμένουμε το 2011. Και δεύτερον, σήμερα είπατε και τονίσατε την πολιτισμική πολυμορφία. Ο αθλητισμός τι ρόλο θα παίξει στις προτάσεις σας, δεδομένου ότι και ο αθλητισμός βοηθάει την πολιτισμική πολυμορφία. Ευχαριστώ κυρία Βασιλείου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο αθλητισμός όντως ήταν το τελευταίο κομμάτι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ήταν και το λιγότερο σημαντικό στην παρουσίασή μου. Μερικές φορές ό,τι αφήνουμε για το τέλος είναι το πιο σημαντικό, γιατί ακριβώς με αυτό ε, δημιουργούνται εντυπώσεις, είναι το κλείσιμο. Και το ήθελα αυτό. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι θα δώσω πολύ σημασία στον αθλητισμό. Πιστεύω στον αθλητισμό. Το είπα ξανά και ξανά ότι για μένα ο αθλητισμός είναι ένα μέσον για να πετύχουμε πολλά καλά πράγματα. Υγεία, ε, δουλειά ομαδική, εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, πράγματα που θέλουμε να προωθήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι μέρος της πολιτισμικής μας ε, κληρονομιάς βρίσκεται και στον αθλητισμό. Μια που ο αθλητισμός αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής μας παράδοσης. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τον αθλητισμό ε, στις χώρες μας μέσω από διάφορα προγράμματα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να δίνουμε χρήματα για τους ομίλους, όμως να τους στηρίζουμε με προγράμματα, με κατάρτιση προχωρώντας με τέτοιου είδου αθλήματα, με παραδοσιακά και παραπέρα, προωθώντας τα. Περιμένω ιδέες από σας Και περιμένω, αφού έχω τις ιδέες αυτές, να προχωρήσω σε προτάσεις. Κύριε Κέλλη, εντάξει, το σημειώνουμε αυτό. δεν μου είπατε γιατί τις προτάσεις σας τις αφήνετε για το 2011 και όχι για το 2010. Να ξέρετε πάντως ότι πρέπει μάλλον στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο να βάζετε τα πέντε αθλητισμού γιατί δύσκολα θα σας αφήσει κανείς να φτάσετε στο τέλος, η πρόεδρος δηλαδή. Ναι, λοιπόν, το πρόγραμμα για τον αθλητισμό ξεκινάει το 2011, διότι έχουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις για τον αθλητισμό, που ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια και συνεχίζονται και το 2010. Οπότε θα συνεχίσουμε με αυτές τις προπαρασκευαστικές ε, δράσεις το 2010 και βάσει της εμπειρίας μας, κατά τη διάρκεια αυτών των προπαρασκευαστικών δράσεων, μαζί, σε συνεργασία μαζί σας δηλαδή, θα διατυπώσουμε το πρόγραμμά μας για τον αθλητισμό στο μέλλον. Ο κύριος Μάτουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα η αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δυναμική. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η επαγγελματική κατάρτιση οι αλλαγές επαγγέλματος είναι πράγματα μεγάλη σημασία στην Ευρώπη. Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι η διαβίου μάθηση και οι αλλαγέ επαγγελματική δραστηριότητα είναι πράγματα που πρέπει να μείνουν στο σημερινό σύστημα εκπαίδευση ή σε ένα άλλο σύστημα που δεχειριζόμαστε με το Υπουργείο εργασία με ή χωρί την εργοδοσία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι ανάγκες που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Η κατάρτιση σίγουρα είναι κάτι αναγκαίο. Έτσι κι αλλιώς. Όπως είπα και πριν, οι ανάγκες σε κατάρτιση και εκπαίδευση αλλάζουν γιατί έχουμε εξελίξει στην τεχνολογία, έχουμε αλλαγές στις αγορές που γίνονται πιο ανταγωνιστικές που χρειάζονται περισσότερες δεξιότητες. Άρα κάθε χώρα μέλος έχει διαφορετικές ανάγκες. Όμως θα έχουμε συνεργασία μεταξύ μας για να δούμε, ακόμα και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τη γνώση που θα συγκεντρώσουμε και πώς θα συνδυάσουμε καλύτερα την εκπαίδευση με την εργασία. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί γιατί είναι αναγκαίο. Αυτό που είναι ξεκάθαρο για όλους σήμερα είναι ότι όσο περισσότερες δεξιότητες, όσο περισσότερα προσόντα έχει κανείς, τόσο περισσότερες εγγύησεις έχει ότι δεν θα βρεθεί στην ανεργία. Αυτή είναι η εμπειρία που πήραμε από την τελευταία κρίση. Αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση είναι οι νέοι με τα λιγότερα προσόντα πέρασε ο καιρός όπου ε, τα άτομα με λίγες δεξιότητες και χαμηλά προσόντα έβρισκαν εύκολα δουλειά. Όχι. Η... Τα υψηλά προσόντα και ιδιαίτερες ε, δεξιότητες είναι αυτές που θα χρειαστούν περισσότερο στο μέλλον. Άλλη ερώτηση κύριε Μάτουλα. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να προσθέσω, μάλλον να ρωτήσω την κυρία Βασιλείου το εξής τι ρόλο θέλει να έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα υπάρξει χώρος για ένα σύστημα παράλληλο ιδιωτικής ε, κατάρτισης από ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή, και τι κινδύνους βλέπει σε κάτι τέτοιο. Για αυτά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο οι εργοδότες, αλλά και τα συνδικάτα των εργαζομένων να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, τη γνώμη τους, τις ανάγκες τους, να υπάρχει δηλαδή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των Ινστιτούτων επαγγελματική Κατάρτισης και του κόσμου των επιχειρήσεων, εργοδοτών και συνδικάτων, κοινωνικών εταίρων δηλαδή. Ευχαριστούμε. Τώρα τα μέλη των Επιτροπών Απασχόλησης και Πρώτα απ' όλα ο κύριος Σόγκορ. Yeah, the lifelong learning program which... Το πρόγραμμα ισόβιας εκ, ε, εκμάθησης είναι ένα πολύ ευρύ πρόγραμμα. Θεωρείται ότι ο προπολογισμό του αρκεί για να καλύψει τα 7 διαφορετικά προγράμματα που υπάρχουν και να επιτρέψει 33 συμμετέχουσες χώρες τη δυνατότητα να υποφεληθούν από το πρόγραμμα. Και μια δεύτερη ερώτηση, πώς θα φροντίσετε ότι θα υπάρξει μηχανισμός ποιότητας του ελέγχου και καλή ισορροπία μεταξύ των συμμετέχουσών χωρών, προκειμένου να δημιουργηθεί επίσης ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα τέτοιο μηχανισμό. Είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα, γιατί όπως είδαμε στο πρόσφατο γλωσσικό θέμα για τη Σλοβακία, και τι γίνεται με τις στατιστικές, το σύστημα στατιστικών πληροφοριών που δίνει πληροφορίες για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος, η κυρία Βασιλείου. Οι προπολογισμοί ποτέ δεν είναι επαρκείς. Και σε αυτό το πρόγραμμα διαβίου εκμάθησης, lifelong learning, ένα από τα, προγράμμα, ένα τα προβλήματα που δεν προβλέψαμε το, την αύξησή του, όπως με το έρεσμο που ελπίζαμε ότι το 2012 θα είχαμε 3 εκατομμύρια φοιτητές συμμετέχοντες δεν θα το φτάσουμε το στόχο αυτό. Και ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια. Σωστά όμως είπατε, είναι και το θέμα της ποιότητας. Σας θυμίζω ότι η ποιότητα είναι και αυτή τη μήμα της χάρτας που υπογράφεται με τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν πρέπει να μας διασφαλίσουν για την καλή ποιότητα των προγραμμάτων. Δική μας ευθύνη είναι αυτές οι διαβεβαιώσεις να υλοποιούνται. Η ποιότητα λοιπόν είναι σημαντική. Ο προπολογισμό είναι σημαντικός. Θα πρέπει όμως να ενθαρρύνουμε και τις κυβερνήσεις, τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία να επενδύσουν στα προγράμματα αυτά και αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειών και των πανεπιστημίων είναι σημαντική για τις ε, καλύτερες περαιτέρω εξελίξεις του συστήματος. Ο κύριος Σόγκορ δευτερολογεί. Τη δεύτερη ερώτηση που σκόπευα να κάνω την υπέβαλε ο συνάδελφος κύριος Σμίτς αφορούσε την προστασία των μειονοτικών γλωσσών. Και απαντήσατε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, βέβαια δεν έχει αυτό και σχέση με την απασχόληση. Η κυρία Ράπτη. Απασχόληση. Είναι παρούσα. Thank you, Mr. President. κυρία Βασιλείου, καλώς ήρθατε θα σας βάλω στην πρόκληση να υποστηρίξετε την πολυγλωσία και τη χρήση της στην πράξη, απαντώντας μου αν θέλετε στη δική σας γλώσσα και τη δική μου. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την παροχή κατάρτισης και διαβίου εκπαίδευσης προκειμένου να παρασχεθούν οι ειδικότητε για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Μιλάω βέβαια για τις πράσινες θέσεις εργασίας θα υποστηρίξετε ισχυρότερες πολιτικές και δημοσιονομικά μέσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους μας να πάρουν τις ειδικότητε που χρειάζονται και νομίζω ότι η οργάνωση μας στη Θεσσαλονίκη κάνει μια πολύ καλή δουλειά η ε, μια πολύ καλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα και προσβλέπουμε στις ε, μελέτες τις οποίες άρχισε ήδη να κάνει για τις ανάγκες της εργασίας στο μέλλον. Θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ε, εμπειρίες και τα στοιχεία τα οποία θα μας δώσουν για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στους νέους να πάρουν εκείνη την εξειδίκευση που θα τους επιτρέψει να βρουν εργασία. Και πρέπει να πω ότι ε, ήταν πραγματικά λυπηρό να δω ότι η χώρα σας είναι μια από τις χώρες που 80% των αποφύτων των πανεπιστημίων είναι άνεργοι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε πού οφείλεται αυτό. Και ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Και να δώσουμε ακριβώς τι ειδικεύσει που χρειάζονται οι νέοι για να μπορέσουν και τι δεξιότητε, Διότι απλά το να τελειώσεις ένα πανεπιστήμιο χωρί να έχει εξειδικευμένε γνώσει και ε, εμπειρίε, δεν είναι αρκετό. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στο να δώσουμε αυτέ τι ευκαιρίε στους νέου μα. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα να το κάνουμε, μέσω των προγραμμάτων μα φυσικά, και θα ενθάρρυνα πάρα πολύ την Ελλάδα να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί τα προγράμματα τα οποία έχουμε, αλλά φυσικά ε, είναι και θέμα ε, λεφτών. Μέσα στα πλαίσια του, ε, των δυνατοτήτων μας, των οικονομικών μας δυνατοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά και της Ελλάδας, να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα προγράμματα που θα βοηθήσουν τους νέους μας. Μπορώ να συνεχίσω για μια δεύτερη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, πολύ σωστά μιλήσατε και συμφωνώ μαζί σας για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ΣΕΝΤΕΦΟ που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και βέβαια υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Κατά τη γνώμη σας, πώς βλέπετε, πώς θα μπορέσετε να συντονίσετε τη δραστηριότητα αυτών των τριών οργανισμών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια κοινωνία της γνώσης ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς. Και θα ήθελα, αν μπορείτε να μου πείτε πιο συγκεκριμένα, αν έχετε στο μυαλό σας, τι θα προτείνετε ώστε αυτή η συνεργασία να γίνει αποτελεσματική, να περπατήσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία. Είναι κάτι διαφορετικό. Εκείνο το Ινστιτούτο είναι ε, ενό πολύ υψηλού επίπεδου Ινστιτούτων το οποίο θέλει να δέσει μεταξύ του την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Έχει μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Συγγνώμη που διακόπτω, επειδή μιλήσατε προηγουμένως για την ανάγκη της τεχνολογίας και την εμπλοκή της με την κατάρτιση. Γι' αυτό ακριβώς το προσθέτω και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει συνεργασία. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο πρέπει να γίνει το flagship της, ε, της, ε, της ε, δικής μας ομάδας. Πρέπει να το κάνουμε το flagship της Ευρώπης. Ε, και, θέλω, και θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι θα γίνει, διότι ε, η τελευταία απόφαση του, ε, της επιλογής των προγραμμάτων, των ε, KICS, το λεγόμενα, των, του Ινστιτούτου, ήταν πολύ επιτυχημένη. Έχει καταφέρει να κεντρήσει το ενδιαφέρον μεγάλων κέντρων καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης και, και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχει το ρόλο του. Απλά είπα ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα άλλα δύο με το Ινστιτούτο. Έχουν φυσικά το κάθε έναν το ρόλο του. Και θα τα εκμεταλλευτούμε. Thank you very much. Mrs. please. Χάρκιν, ε, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, σε μία από τις απαντήσεις σας μιλήσατε για τον στόχο που έχετε να προωθήσετε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως ίσως έχετε ακούσει, 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι εθελοντές και η εθελοντική δραστηριότητα είναι κομμάτι της, ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και όπως είπε ο κ. Σκουρία το 2011 έχει οριστεί ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού οπότε στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα πρώτα απ' όλα πως σκοπεύετε να δημιουργήσετε συνέργειες μεταξύ υπαρχόντων προγραμμάτων όπως το νεολαία σε δράση, διαβίου, κατάρτιση κτλ. και τις δραστηριότητε του 2011 και δεύτερον πώς βλέπετε εσείς να συνεισφέρει το ευρωπαϊκό έτος ε, εθελοντισμού στην απασχολησιμότητα των εθελοντών. Ναι, ευχαριστώ. Όπω είπατε, το 2011 είναι έτος εθελοντισμού. Η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Η ε, δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ξεκινήσει ήδη. Λυπούμε για το ότι δεν θα είμαι εγώ η επικεφαλής επίτροπος, αλλά βεβαίως θα συνεργαστώ πλήρως ε, με τους ε, συναδέλφους στον τομέα αυτών και νομίζω πως ο εθελοντισμός θα πρέπει να οφηθεί προς την σωστή κατεύθυνση γιατί φοβάμαι πως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ο εθελοντισμός να αντικατοστήσει ή να δώσει μάλλον την ευκαιρία στους ε, εργοδότες να προσφέρουν εθελοντισμό αντί για αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, ο εθελοντισμός, μια χρήσιμη έννοια, πρέπει να την προωθήσουμε με σκοπό να προωθήσουμε τις εμπειρίες ε, και την γνώση των ανθρώπων, αλλά όχι να, μην αλλά όχι να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση από τους εργοδότες. Κατά διάρκεια λοιπόν αυτού του έτους πρέπει να βρούμε τρόπους να δούμε πώς θα προωθήσουμε τον εθελοντισμό να διατηρηθεί δηλαδή αυτή η ισορροπία μεταξύ αμοιβόμενης και εθελοντικής εργασίας. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση. Ναι, κυρία Χάρκιν. Συμφωνώ πλήρω με την Επιτροπή πώ δεν πρέπει ο εθελοντισμός ε, να αντικαταστήσει την αμοιβόμενη εργασία. Αλλά ε, επειδή πρόκειται ακριβώ για μια άτυπη μορφή μάθησης για πολλούς ε, εθελοντές και πράγματι ενισχύει τις ικανότητές τους και διευκολύνει την επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να το έχετε αυτό κατά νου σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα προτείνετε για συνέργειε μεταξύ ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν. Η κυρία Βασιλείου, έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα για τον εθελοντισμό και έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχή. Και οι μελέτες μας δείχνουν το όφελος της εθελοντικής εργασία όσον αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των εμπειριών. Και Υπάρχει κάτι στο οποίο θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση. Η συνεισφορά του εθελοντισμού στην ε, κοινωνική σφαίρα, στην ανάμιξη των ανθρώπων στη δημόσια ζωή. Τους βοηθάει να αντιληφθούν καλύτερα τις ανάγκες της κοινωνίας, τα ωφέλη της δικής τους προσφοράς στην κοινωνία. Οπότε η κοινωνική πτυχή του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό λέω πως όλα τα προγράμματα σε σχέση με τον εθελοντισμό πρέπει να ενισχυθούν. Ευχαριστώ, κυρία Σρέντερ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βασιλείου, μιλήσατε για το ότι θα αναφερθείτε σε όλες τις ανάγκες ε, του πληθυσμού ε, όσον αφορά την εκπαίδευση, αλλά βεβαίως και των επιχειρήσεων και μιλήσατε για τις ε, νέες δουλειές στην πράσινη οικονομία. Διαπιστώθηκε από μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως θα απαιτηθούν μέτρα επανεκπαίδευσης κυρίως μεγαλύτερων εργαζομένων μεγαλύτερων σε ηλικία ενώ που θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Τι σκοπεύετε να κάνετε, σκοπεύετε να δω, κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις επανεκπαίδευση αυτών των ανθρώπων για να δώσουν και τα κράτη-μέλη ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους ανθρώπους για να εκμεταλλευτούμε και αυτό το δυναμικό και να μην το χαραμίσουμε αλλά να τους επανεντάξουμε στην παραγωγική διαδικασία. Σας ευχαριστώ κυρία Βασιλείου. Ευχαριστώ. Πράγματι, το να δοθεί η δυνατότητα στους ενήλικες να συνεχίζουν τη διαδικασία μάθησης είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό είναι η διαβίου μάθηση. Η διαβίου μάθηση πρέπει να ξεκινάει πριν από το σχολείο ήδη και να συνεχίζει είχαν ένα σύνθημα στις μου που δεν μου άρεσε και πάρα πολύ ε, γιατί λέει μέχρι τον τάφο, εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θα έλεγα μέχρι τον τάφο, ακούγεται έτσι κάπως μακάβριο, ας πούμε και μετά τη συνταξιοδότηση. Πρέπει να είμαστε δραστήριοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Τα προγράμματα λοιπόν διαβίου κατάρτισης δεν αφορούν μόνο τους νέους, αλλά και τους ενήλικες που θέλουν να παραμείνουν δραστήριοι και πρέπει να το ενθαρρύνουμε αυτό γιατί είναι καλό για όλους εγώ που προέρχομαι από τον τομέα της υγείας, μπορώ να σας πω πως μία πολιτική μας ήταν η ενεργή και μεγάλη ζωή. Δηλαδή για να είμαστε ενεργοί σε μεγάλη ηλικία, δείτε μένα δηλαδή, εγώ παραμένω ενεργή γιατί θεωρώ πως έτσι πρέπει και πρέπει να συνεχίσω να μαθαίνω. Οπότε πρέπει αυτές τις δυνατότητες να τις έχουν όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σέντερ, να επανέλθω στην ε, πρωτοβουλία της ε, νεολαίας ε, σε κίνηση. Αλλά εδώ πέρα νομίζω πως δεν υπάρχουν και αρκετά εκπαιδευμένοι νέοι, τι σκοπεύετε να κάνετε στη βασική εκπαίδευση, ειδικά για τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να εκμεταλλευτούμε και αυτά τα ταλέντα. Έχετε συγκεκριμένες ε, ιδέες εδώ πέρα. Παρακαλώ κύριε Βασιλείο Νομίζω πως η ένταξη όλων στα προγράμματά μας είναι πολύ σημαντική και είχα πει πριν πως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στα παιδιά τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία από την οικογένειά τους να κάνουν τα πράγματα τα οποία θέλουν για εκπαίδευση, κατάρτιση, κινητικότητα. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση σε ανθρώπους από αυτές τις κατηγορίες. Και στους μετανάστες βεβαίως και αυτή είναι μέρος της κοινωνίας μας. Οπότε το να ταιριάξουν οι ανάγκες της αγοράς με τις δεξιότητες που δίνουμε στους νέους δεν έχει στόχο μόνο να εξυπηρετήσει την οικονομία αλλά και να προσφέρει καλύτερες προοπτικές στους νέους για μια καλύτερη ζωή. Αυτός είναι ο στόχος ε, όλων των προσπαθειών μας. Να προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή στους ανθρώπους, όποια ηλικία και αν έχουν, όποιο και αν είναι το υπόβαθρό του, ε, όποιε ικανότητε και αν έχουν, γιατί ακόμα και τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες έχουν ικανότητε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τι ικανότητε που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, όσοι δεν ακούνε εδώ πέρα, ε, παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα. Ναι, εκεί ο νεάρο κοκκινομάλης. Είστε εδώ πέρα προσκεκλημένος, ε, δεν είναι εδώ μέρος να κάνετε την κουβέντα σας είναι μια υποψήφια επίτροπος. Εδώ δεν είναι ευγενικό αυτό. Με συγχωρείτε που ξεχωρίζω εσά, εσά είδα εκείνη τη στιγμή. Ο κύριος Higgins, νομίζω απουσιάζει, περνάμε στον κύριο Σιμάνσκι, ούτε αυτός. Ο κύριος Χίρς, νομίζω, η κυρία Χίρς, τον αντικαθιστά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βασιλείου, έχουμε συχνά το πρόβλημα το ότι ειδικά στις ε, θετικές και στις τεχνικές επιστήμες έχουμε μία έλλειψη και στον παιδαγωγικό τομέα υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν έχουμε άντρες π.χ. στην πιαγωγία ή στο δημοτικό σχολείο και από την άλλη βεβαίως ε, ε, λείπουν γυναίκες στον τεχνικό τομέα. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να ε, αντιμετωπίσουμε το ότι η απόφαση του τι θα γίνει κανείς όταν μεγαλώσει, δεν τελευταίες τελευταίε δύο τάξεις σχολείου, αλλά πολύ νωρίτερα. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε για να ενθαρρύνετε τις γυναίκες, τα κορίτσια μάλλον, ήδη από νωρίς να α, κατευθυνθούν προς τον τεχνικό τομέα, αλλά και οι άντρες να μην διαλέγουν μόνο τα λεγόμενα κλασικά αντρικά επαγγέλματα. Η κυρία Βασιλείου, ευχαριστώ. Θίξατε ένα ζήτημα το οποίο μου είναι ιδιαίτερα αγαπητό, την ισότητα των φίλων. Και νομίζω ξεκινά από την οικογένεια. Η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνουν τους νέους τα κορίτσια ή τα αγόρια να κατευθυνθούν τα κορίτσια προς τις θετικέ επιστήμες ή τα αγόρια να γίνουν δάσκαλοι. Στη χώρα μου 95% των διδασκόντων είναι γυναίκες. Και δεν είναι υγιές αυτό. Βεβαίως να δουλεύουν οι γυναίκες. Αλλά τα παιδιά πρέπει να έχουν και την εμπειρία και των δύο φίλων. Πρέπει να υπάρχει ισότητα σε όλα τα επαγγέλματα. Και η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην ενθάρρυνση των παιδιών ε, στο τι θα κάνουν στη ζωή τους. Αλλά και εμείς έχουμε ρόλο να παίξουμε. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να προσπαθήσουν. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ καλό α, ε, υπόδειγμα. Δηλαδή να στέλνουμε τα παιδιά όταν είναι στο σχολείο να δουν πώς είναι τα διάφορα επαγγέλματα. Γιατί όταν είναι κάποιος 16-17 δεν ξέρει τι σημαίνει νομικά, τι είναι η οικονομία ή τι είναι οι κατασκευές ή η διδασκαλία. Πρέπει να το δοκιμάσουν, πρέπει να το δουν, να πάνε να δουν από κοντά και να κρίνουν από μόνο τους αν τους αρέσει. Αλλά συνήθως φοβάμαι οι μητέρες λένε στις κόρες τους «Α, θα γίνεις καλή δασκάλα». Και στα αγόρια λένε «Θα γινώσουν καλός υδραυλικός». Οι ερευνητέ. οχι μπορουν να γινουν Μπρούτλαντ ήταν ε, πρωθυπουργό της Νορβηγία, ένας ε, δάσκαλος, ένας μαθητής αγοράκι είχε ρωτήσει τον την δασκάλα «Κυρία, μπορώ και εγώ να γίνω πρωθυπουργό, γιατί εδώ και τα πρότυπα είναι πάρα πολύ σημαντικά». Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Ε, έχετε συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Χίρις. Ναι, μία ερώτηση ακόμα, κάπως πιο εξειδικευμένη. Ένα θέμα το οποίο θα αποτελέσει πρόκληση και για εσάς. Έχουμε μία χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρει συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην Ευρώπη έχουμε πάρα, πολλούς, ε, πάρα πολλά παιδιά, νέους που είναι παιδιά παρανόμων μεταναστών. Πώς θα διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Βλέπετε εδώ πέρα την ε, δυνατότητα συνεργασίας με άλλους ε, συναδέλφους σας ε, στην Επιτροπή για να βρείτε τις δυνατότητες εντός των κρατών μελών να διασφαλιστεί αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα και αυτών των παιδιών. Σας ευχαριστώ κυρία Βασιλείου. Νομίζω πως το οφείλουμε σε όλα τα παιδιά να έχουμε σωστή να έχουν σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση. Και αυτό βεβαίως είναι, περιέχεται και στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την οποία έχουμε όλοι κυρώσει. Οπότε πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Γνωρίζω πως ε, η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την κοινωνική τους ε, πολιτική, ανάλογα με τις ε, οικονομικές ανάγκες του κάθε κράτους, αλλά είναι κάτι που πρέπει να ενθαρρύνουμε, είναι ανθρώπινο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Σας ευχαριστώ. κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Ψήφα Επίδροε. επειδή είμαι πανεπιστημικός καθηγητής, έχω διατελέσει, θα αναφερθώ στη διαδικασία της Μπολόνια και στην, ε, τα σχετικά. Μέχρι στιγμή η πολιτική εφαρμόστηκε επιτυχώ όσον αφορά τις, την ανώτατη εκπαίδευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες μέλη. Θεωρείται αυτή την ε, κίνηση επιτυχία ή κατά τη γνώμη σας χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση προκειμένου να ληφθούν υπόψη η κατα τη γνωμη χρειαζεται αναγνώριση πτυχίων, και η μετανάστευση κατά κάποιο τρόπο των φοιτητών μεταξύ των διαφόρων πανεπιστημίων. Η κυρία Βασιλείου. Θεωρώ τη διαδικασία Μπολόνια ως επιτυχία. Είναι success story όπως είπατε κι εσείς. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο πέρας αυτής της διαδικασίας. Όπως είπα και πριν, σύντομα θα γιορτάσουμε τα 10 χρόνια γενέθλια της ε, διαδικασίας Μπολόνια. Πρέπει να ανανεώσουμε την δέσμευσή μας, την υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε. Έχουμε πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό στη σύγκληση των πανεπιστημίων σε πολλά θέματα. Από την άλλη μεριά έχουμε το θέμα της ποιότητας, την ταξινόμηση όσον αφορά τα πανεπιστήμια, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, την αυτονομία των πανεπιστημίων. Όλα αυτά είναι εξίσου σημαντικά και θα πρέπει να τα ε, αντιμετωπίσουμε από εδώ και μπρος δευτερολογία του κυρίου Μεζάρος. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, πώς αξιολογείται το έργο λίγων ετών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Θεωρείται γενικά ότι το να υπάρξουν κοινά Ινστιτούτα στην Ευρώπη ενσωματώντας τα ευρωπαϊκά μυαλά με την έρευνα και την ανάπτυξη είναι ένας καλός τρόπος για να πετύχουμε αριστεία. Η απάντησή μου είναι ένα μεγάλο ναι. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας που μόλις τώρα άρχισε να δουλεύει είναι ένα άριστο μοντέλο ένωσης του τριγώνου. Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη. Εκπαίδευση. Πετύχαμε σωστά την έναρξη. Το φθινόπωρο θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Θα έχουμε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το φθινόπωρο. Και υπάρχει και κάτι άλλο που με ευχαριστεί. Ένας από τους στόχους μας ήταν να ελκύσουμε ανθρώπους από τη βιομηχανία για να κλείσει το, το τρίγωνο και το πετύχαμε. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις πήραν μέρος στο διαγωνισμό, στη διαδικασία. Επίσης είχαμε καλή συμμετοχή και από τις νέες χώρες μέγη της Κεντροανατολικής Ευρώπης. Ουγγαρία, Πολωνία. Ε, ήταν επιτυχία λοιπόν. Ο κύριος Εντσιού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βασιλείου, σας συγχαίρω για το ότι είστε η υποψήφια επίτροπος και ελπίζω και σας εύχομαι όλα τα προγράμματά σας να υλοποιηθούν στη διάρκεια της θητείας σας. Θα αναφερθώ στην ψηφιακή τεχνολογία, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά κονδύλια. Και θα ήθελα να μας πείτε Πώς θα υποστηρίξετε αυτό το πρόγραμμα ως βάση της ψηφιακής τεχνολογίας και ως θύρα για τις βιβλιοθήκες, όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα. Θύρα εισόδου, πόρταλ. Άλλες ιστοσεγγίδες θα μπορούσαν να δώσουν τις πληροφορίες που οι πολίτες, για τις οποίες οι πολίτες πρέπει να πληρώνουν. Απάντηση. Η ψηφιακή κοινωνία είναι εδώ και πρέπει να υποστηρίξουμε τη δουλειά που γίνεται στον τομέα αυτό. Αλλά πρέπει να από την άλλη μεριά να κατανοούμε ότι ας πούμε ότι υποστηρίζουμε χίλια προγράμματα. Μελετάω το χαρτοφυλάκι αυτό εδώ και τέσσερις εβδομάδες το πολύ. Δώστε μου χρόνο να εξοικειωθώ με όλα τα προγράμματα αυτά Δυστυχώς δεν τα γνωρίζω όλα. Αυτό που αναφέρετε δεν το γνωρίζω. Πάντως σας διαβεβαιώνω ότι θα μάθω περισσότερα, θα επανέλθω στο θέμα αυτό για να σας απαντήσω. Δευτερολογία του κυρίου Έντσιου. Αν η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη η ε, γίνει βάση δεδομένων, θα συμφωνούσατε να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου αυτής της ψηφιακής βιβλιοθήκης για τα εκπαιδευτικά όργανα, πολιτιστικούς, πολιτιστικά όργανα κλπ. Διότι όλοι ξέρουμε ότι οι φοιτητέ, οι ερευνητέ, οι καθηγητές είναι εγγύηση για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης. Επειδή όμως τα πνευματικά δικαιώματα είναι εμπόδιο στην πρόσβαση, τι θα κάνετε. Απάντηση. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο που αναφέρεται, τα copyright, τα πνευματικά δικαιώματα. Το είπα και στην αρχή. Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αμείβονται σωστά για το έργο τους. Άρα το copyright δεν τίθεται ένα αμφιβόλο. Αν να πληρώνουμε πνευματικά δικαιώματα λοιπόν, θα δούμε πού, όπου γίνεται, να προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στον κόσμο. Και αν προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στους Ευρωπαίους πολίτες, τι θα γίνει με τους πολίτες άλλων χωρών του πλανήτη που θα ήθελαν και αυτοί να επωφεληθούν από τη σύστημα. Θα ήταν άνηση μεταχείριση. Μάλλον κάτι τέτοιο. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό που θα κάνουμε είναι θα το μελετήσουμε. Καταρχήν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα και χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη να ολοκληρωθεί. Και μετά θα δούμε αν μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Πρόεδρος. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω στον ε, κύριο Εντσίου πως ε, το Ευρωπαϊκό είναι στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Κρούς. Γιόρνταν Τσίσελη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλείου. Έχω μια ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Με ακούτε? Με ακούγομαι τώρα? Ωραία. Ξεκινάω και πάλι. Επαναλαμβάνω, έχω μια ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, παρακαλώ. Το Ινστιτούτο αυτό είναι δικιά σας αρμοδιότητα και έχει να κάνει με την έρευνα και την καινοτομία που όμως αποτελούν αντικείμενο άλλου επιτρόπου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς θα διασφαλίσετε τα μέτρα που λαμβάνονται για το Ινστιτούτο να συντονίζονται με τα μέτρα που παίρνουν άλλοι επίτροποι. Θέλουμε μια οικονομία με καινοτομία. Εσείς θα σεβαστείτε τη συμπερίληψη των επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο αυτό. Θα διασφαλίσετε δηλαδή ότι η δουλειά του Ινστιτούτου θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των επιχειρήσεων. Και τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου το Ινστιτούτο αυτό να μην γίνει ένα κέντρο καθαρά διοικητικό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βασιλείου. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ο Επίτροπος Μπαρόσο θέλει πάρα πολύ να προωθήσει το Ινστιτούτο αυτό, ώστε να στεφθεί με επιτυχία. Και ξέρω ότι όλοι οι επίτροποι θέλουν να συνεργαστούμε όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να πετύχει το Ινστιτούτο αυτό. Δεύτερον, δεν έχω αμφιβολία, έχοντας ήδη συναντηθεί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου του Ινστιτούτου αυτού, για το ότι πρόκειται για ένα άτομο μεγάλης αποφασιστικότητας και πρόκειται για έναν οραματιστή με πολλή εμπειρία σε αυτό το τομέα. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα πετύχει το Ινστιτούτο. Άκουσα, δεν έχω βέβαια συναντηθεί ακόμα μαζί του, αλλά ξέρω ότι έχουμε και ένα πολύ καλό διευθυντή που έχει ήδη αναλάβει τα καθήκοντά του στη Βουδαπέστη. Πολύ σύντομα το Ινστιτούτο νομίζω την Άνοιξη θα λειτουργεί πλήρως και θα είναι πλήρως αυτόνομο και ανεξάρτητο. Κατόπιν τούτου και όταν ξεκινήσει η δουλειά, μία ευθύνη έχουμε. Και εδώ είναι δηλαδή που μπορεί να βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο και θα συνεργαστούμε και είμαι βεβαία ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέλει, προκειμένου να περάσει το μήνυμα του Ινστιτούτου στην εκπαιδευτική κοινότητα, την ερευνητική κοινότητα και την κοινότητα της καινοτομίας. Γιατί θέλουμε να αποτελέσει μια αναβαρχίδα το Ινστιτούτο αυτό. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Στην προηγούμενη θητεία εγώ το στήριξα αυτό το σχέδιο και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα συνεργαστούμε με επιτυχία πάνω σε αυτό. Θα πετύχουμε το τρίγωνο αυτό της γνώσης στο οποίο αναφερθήκατε. Μία όμως επιπλέον ερώτηση παρακαλώ όσον αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι και η αδυναμία του τριγώνου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τι άποψη έχετε από αυτού. Πώς πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορέσουν να συνεργαστούν με το Ινστιτούτο αυτό καλύτερα, προκειμένου η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της οικονομίας μας. Η κυρία Βασιλείου. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδούμε την αξιολόγηση των ε, εκπαιδευτικών ιδραμάτων. Σίγουρα έχουμε πολλούς ειδικού εδώ, αλλά εγώ πιστεύω ότι περισσότερο Περισσότερο από την ταξινόμηση αυτή που έχει γίνει των πανεπιστημίων βασίζεται στην έρευνα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλους παράγοντες και άλλα κριτήρια για να αξιολογήσουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για παράδειγμα, τρόπος διδασκαλίας. Ε, πόσο διεθνή είναι τα ιδρύματα αυτά. Πόσο κοντά βρίσκονται στην ε, κοινότητα, στον κόσμο. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να εξυγχρονίσουμε τα πανεπιστήμια μας. Θέλουμε τα πανεπιστήμια μας να λειτουργούν καλύτερα και να δίνουν την ευκαιρία στους νέους να μπορούν να κάνουν τις σωστές επιλογές. Πρέπει να είναι αυτό αποστολή των πανεπιστημίων, ώστε οι νέοι να μπορούν καλύτερα να πάρουν την απόφαση τι θα σπουδάσουν, πού θα το σπουδάσουν. Αυτό θα ενισχύσει πιστεύω τα πανεπιστήμια μας στην Ευρώπη και θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά και από τα καλύτερα του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος, πήγαμε πολύ γρήγορα. Και έτσι μας έχει περισσέψει χρόνος. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω το σύστημα Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο σε πέντε. Μία ερώτηση, μία απάντηση χωρίς συμπληρωματική ερώτηση. Κυρία Χάιμ, η κυρία Καμερεβεδό, Άρης, Βάτιμο, Σάρκινς και Φίσα. Αυτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Βασιλείου. Πολλά από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε είναι σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Και εκεί πέρα λαμβάνονται οι πρωτοβουλίες. Το τοπικό επίπεδο ενισχύεται με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Τι άποψη έχετε για μια πιο ενισχυμένη και δοδημημένη συμμετοχή των τοπικών αρχών όσον αφορά και την σύλληψη και την εφαρμογή των προγραμμάτων πολιτισμού, εκπαίδευση και αθλητισμού και πώ θα διασφαλίσετε την έγκαιρη εμπλοκή του, παραδείγματο χάρη μέσω πρωτοβολιών και δράσεων στον ε, τομέα του εθελοντισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμπλέξουμε ακόμη περισσότερο του ανθρώπου επιτόπου. Ναι. Νομίζω πως ε, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, όλες οι πτυχές του χαρτοφυλακίου μου, ο αθλητισμός, είναι θέματα τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να κινητοποιήσουμε και να αναζητήσουμε στήριξη από τα κράτη-μέλη οπωσδήποτε, αλλά και από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πλεονέκτημα ποιο είναι, γιατί από τις μελέτες που κάναμε είναι σαφές πως όταν οι ε, τοπικές αρχές δίνουν βάρος σε έργα όπως τα δικά μας, εποφελούνται. Και χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα πως ε, προσεκλήθη η αρμόδια Γενική Διεύθυνση φέτος για πρώτη φορά να λάβει μέρος ε, στη σχετική εκδήλωση που οργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βασιλείου, θα επανέλθω στον τομέα του πολιτισμού και συγκεκριμένα των οπτικοακουστικών μέσων που αποτελούν σημαντικό τμήμα του πολιτισμού στην ε, κοινωνία μας και από πλευράς ε, του ανταγωνισμού, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό η ερώτησή μου συμφωνείτε πως ιδιαίτερα τα δημόσια ΜΜΕ αποτελούν ισχυρές εγγυήσεις για τον πλουραλισμό και την πολιτισμική πολυμορφία και αν ναι, ποια στήριξη μπορείτε να μας πείτε ότι θα δώσετε εσείς στο πλαίσιο βέβαια πάντα των αρμοδιοτήτων της ε, Κομισιόν για την περαιτέρω ανάπτυξη των δημοσίων ε, ραδιο-τηλεοράσεων στην Ευρώπη. Νομίζω πως είναι ένας πολύ σημαντικός ε, τομέας ειδικά όσον αφορά την πολιτισμική πτυχή των οπτικοακουστικών μέσων, λέει η κυρία Κάμερφερτ. Κυρία Βασιλείου, συμφωνώ πως δεν θα πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση των ΜΜΕ και τα δημόσια ΜΜΕ βεβαίως θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο γιατί έχουν σαφώς ρόλο να παίξουν και πρέπει να τον επιτελούν αυτόν σωστά, να ενημερώνουν το κοινό, να ενθαρρύνουν τον πολιτισμό, τον διαπολιτισμικό διάλογο. Όλα αυτά δεν προβάλλονται τόσο από τα ιδιωτικά μημεία γιατί έχουν άλλα συμφέροντα, έχουν ιδιώτες επενδυτές και τα συμφέροντά τους. Αλλά πρέπει να αντιληφθείτε βεβαίως πως η Κομισιόν δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Εμείς μπορούμε να δείξουμε το ενδιαφέρον μας και να ενθαρρύνουμε, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τον ρόλο που πρέπει να παίξουν. Ευχαριστώ, Μπορείς. Για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Αν, θέλετε Αν θέλουμε να έχουμε μια δυναμική οικονομία, δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει αν δεν έχουμε καλό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης με καινοτομίες. Η υποψήφια για θέματα καινοτομιών αναφέρθηκε σε μια ομάδα επιτρόπων που θα είναι αρμόδιοι. Γι' αυτό εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι τα κονδύλια που θα πάνε στην έρευνα και την ανάπτυξη θα βοηθήσουν και την κατάρτιση Πάμε προγράμματα ε, για ε, θύρες εισόδου στο ίντερνετ κλπ. Γενικά για την εκπαίδευση, για την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τους διδάσκοντες. Όταν αναφέρθηκα στο όραμά μας για το μέλλον, για εκπαίδευση, κατάρτιση, δεξιότητες κλπ. Και είπα ότι δεν εννοούμε μόνο τα πανεπιστήμια, την τυπική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι μια προσπάθεια εγκάρσια που προσπαθεί να δώσει στους ανθρώπους τις καλύτερες δυνατές δεξιότητες για να επιζήσουν, να έχουν μια καλή ζωή στους καιρούς που ζούμε με τις τόσες προκλήσεις και ο πρόεδρος Μπαρόσο δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση με την ευρία έννοια του όρου και την ενίσχυση αυτού του τριγώνου γνώσης, εκπαίδευση, καινοτομία, έρευνα και εγώ όσο μπορώ θα υποστηρίξω την προσπάθεια να υπάρχουν επαρκή κονδύλια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάτιμο. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω σε αυτό που είπατε πριν για τα οπτικοακουστικά. Εφιστώ την προσοχή της υποψήφιας επιτρόπου στο εξή. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς τον υπόλοιπο κόσμο, ένα, το πρώτο θα έλεγα είναι πολιτιστικά προϊόντα, μουσική, βίντεο, ταινίες κλπ. Σήμερα μιλήσαμε πολύ για κατάρτιση, εκπαίδευση και σχολεία, αλλά εδώ για την ευρωπαϊκή κουλτούρα η οποία απορροφάει πολιτιστικά προϊόντα ετερογενή πολλές φορές με ιδεολογικές συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έθεσε το ερώτημα. Δεν έχω, δεν έχω απάντηση. Σας το θέτω ως ερώτημα. Σκεφτείτε το. Κυρία Βασιλείο, όντως το πρόγραμμα για τα νέα μίντια, το νέο πρόγραμμα αυτό, που συνδέεται με το χαρτοφυλάκιό μου, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε όσο πιο καλά γίνεται. Ειλικρινά, δεν θεωρώ ότι έχω τα επαρκή κονδύλια στα χέρια μου για αυτό το μεγάλο έργο. Διότι ο τομέας των οπτικοακουστικών, η ποιότητά του και πιστεύουμε ότι θέλουμε να προωθηθεί καλής ποιότητας οπτικοακουστικό προϊόν, χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. Αν δούμε το τι κονδύλια έχουμε σήμερα, λαμβανωμένο υπόψη του λαβρωμένης υπόψη της σημασίας του έργου πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα ακόμη. Έχουμε ένα νέο σχέδιο να δοθούν εγγυήσει στις εταιρείε που παράγουν τα προϊόντα αυτά ιδιαίτερα στην εποχή των πιστοτικής πίεσης και στενότητας που ζούμε γιατί οι τράπεζες δεν είναι εύκολα πιστώσεις στον οπτικό ακουστικό τομέα. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εγγύησεων για να τους βοηθήσουμε. Αν δούμε όμως το ποσό των χρημάτων, τα νούμερα, δεν αρκεί. Πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα, πρόεδρος. Ο κύριος Φίσερ. Ευχαριστώ. Στην επιστολή του κυρίου Μπαρόσο στο τρίτο σημείο αναφέρεται στην κινητικότητα όσον αφορά την εμπειρία σε θέματα διδασκαλίας είναι πιο εύκολο να εγγυθούμε την κινητικότητα των φοιτητών. Των διδασκόντων όμως πώς θα την εγγυθούμε. Εδώ στην προηγούμενη θητή ακούσαμε τόσα πολλά για τον Πολωνό υδραυλικό που πάει και δουλεύει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ένας καθηγητής ένας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου πώς μπορεί να πάει στο Πανεπιστήμιο μιας άλλης χώρας, αυτό πώς θα το βελτιώσετε. Κύριε Βασιλείου, ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικό οι διδάσκοντες να έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους μας. Η κινητικότητα των καθηγητών. Πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα γι' αυτό όμως. Ακριβώς γιατί γνωρίζουμε ότι οι διδάσκοντες εκτός από τη δουλειά τους έχουν τις οικογένειές τους και δυσκολεύονται να τις αφήσουν για να πάνε αλλού. Στο πρόγραμμα Marie Curie υπάρχει όμως ένας ελαστικός στόχος, προκειμένου οι ερευνητές που συμμετέχουν να μπορούν καλά να συνδυάσουν την οικογενειακή του ζωή με την μετακίνηση. Πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει για να ευνοήσουμε και να ενισχύσουμε την κινητικότητα αυτή μεταξύ των διδασκόντων. Είναι ένα αγώνα που αξίζει τον κόπο πάντω. Ο κύριος Τέρκη την τελευταία. Αλλά μην μα μιλήσετε για την ουγγρική γλώσσα πάλι, μα το λέτε αυτό κάθε φορά. Για την υποψήφια επίτροπο. Όντω 70% των εδαφών τη έχασε η Ουγγαρία και σήμερα 3 εκατομμύρια Ούγγροι ζουν σε γειτονικέ με την Ουγγαρία χώρες, όπου η ουγγρική κοινότητα αντιμετωπίζει περιορισμούς όσον αφορά την άσκηση του γλουσικού της δικαιώματος και του πολιτιστικού της δικαιώματος με τη συνθήκη του Τριανών πριν από 90 χρόνια λοιπόν. Εσείς προσωπικά πώς θα φροντίσετε η ευρωπαϊκή πολιτική να είναι τέτοια που να μην μπορεί να υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση σε βάρος ορισμένων Ευρωπαίων πολιτών, αλλά αντίθετα να προωθούνται οι μειονοτικές γλώσσες βάσει του πνεύματος της Ευρώπης που είναι υπέρ της ενίσχυσης της πολιτισμικής πολυμορφίας. Σας ευχαριστώ. Δεν θα σας απαντήσει η κυρία Βασιλείου σε αυτό. Απάντησε τρεις φορές ήδη, νομίζω ήταν ικανοποιητικέ. Οι απαντήσεις πρέπει να τελειώσουμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πειθαρχία που επέδειξαν και την κυρία υποψήφια επίτροπο. Κυρία Βασιλείου, θα σας δώσω ακόμη μία φορά το λόγο για να κάνετε μία σύντομη δήλωση για να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you, ε, Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις ερωτήσεις σας και για την τόσο ζωντανή και καρποφόρα συζήτηση που είχαμε. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα είναι χαμένος χρόνος. Είναι κάτι το οποίο εμπλουτίζει τη δικιά μου εμπειρία και το οποίο θα θυμάμαι προκειμένου να συνεχίσω το έργο μου εφόσον επιβεβαιωθεί ο ορισμός μου στη θέση της Επιτρόπου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι πολύ σημαντικές. Με το νέο πλαίσιο που έχουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας και βάσει των αρχών που έχει καθορίσει με τις κατευθυντήριες γραμμές του ο κ. Βαρόσο για τη νέα εντολή της Επιτροπής, είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να επενδύσουμε προσεκτικά και αποτελεσματικά σε θέματα κλειδί προκειμένου να επηρεάσουμε τη ζωή όλων των Ευρωπαίων προς το καλύτερο σήμερα αλλά και ακόμα περισσότερο αύριο. Θυμάμαι πολύ καλά τα σχόλια που έκανε ένας από τους αξιότιμους ευρωβουλευτές εδώ, μιλώντας για κατασπάληση δημοσίου χρήματος. Σας διαβεβαιώ ότι όσον αφορά τη δικιά μου τη δουλειά, ό,τι αποφασίζουμε και ό,τι κάνουμε θα έχει θετικές επιπτώσεις πάνω στις ζωές των πολιτών μας και δεν θα σπαταλάμε χρήμα. Πρέπει να επενδύσουμε πρώτα απ' όλα στην νεολαία προκειμένου να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχουν για το μέλλον. Πρέπει να ενισχύσουμε την, την ε, κοινωνία της γνώσης. Πρέπει να φροντίσουμε για την διαβίου εκμάθηση, προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι για το μέλλον. Να φροντίσουμε για βιώσιμη πολιτιστική βιομηχανία, προκειμένου να ενισχύσουμε και τη γνώση αλλά να φροντίσουμε και για καλές αμοιβέ απέναντι στους δημιουργούς μας. Να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, να την προωθήσουμε επίσης και να βρούμε νέους τρόπους προκειμένου ο αθλητισμός να στηριχθεί ακόμα περισσότερο ως μέσο που βελτιώνει τη ζωή των Ευρωπαίων. Και δεν είναι τυχαίο που ο αθλητισμός προστέθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας ως ένας από τους στόχους μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε, για την εμπειρία αυτή. Όπως είπα και στην αρχή, είναι η έκφραση της δημοκρατίας αυτές οι ακροάσεις. Και χάρηκα πάρα πολύ που συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία. Να ξέρετε ότι εκτιμά όλος ιδιαίτερος τη συνεργασία που έχω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εσά όλος ιδιαίτερος, και θα προσπαθήσω να κερδίσω κι εγώ από τη δικιά σας εμπειρία, μακρά εμπειρία που έχετε ορισμένη από εσά, προκειμένου να ε, τα βγάλω πέρα ακόμα καλύτερα με το χαρτοφυλάκιο που με τίμησε ο πρόεδρος Βαρός, εφόσον βέβαια επιβεβαιωθεί ο ορισμός μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ, κύριε υποψήφια. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουμε απόψε, αλλά μπορώ να σας πω πως ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία μας σήμερα και πραγματικά επιδείξατε πάρα πολύ μεγάλη δέσμευση για αυτούς τους τομείς που μας απασχολούν και ελπίζω αυτό να διαρκέσει. Να πω τώρα εδώ πέρα στους συναδέλφους, στους συντονιστές, πως απόψε 8 η ώρα συνεδριάζουμε στο 1G3